Okay, friends, we'll start Αρχίζουμε τη ψηφοφορία, αγαπητοί. Σε λίγα λεπτά, παρακαλώ, καθίστε. Και ετοιμάστε τις ηλεκτρονικές κάρτες. Βάλτε τις στη συσκευή μπροστά σας. Είστε έτοιμοι. 14. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ. Those against. Abstentions. Απο, κατά αποχές. You all voted. Yeah. Okay, we'll take an electronic vote in favor. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Υπέρ. Πρόκειται τα χρήματα του Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση, αλλά θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Έτοιμοι. Πέρας. Υπόθεση Fiat Auto Poland. 43-3. Το επόμενο. Ταμείο την Παγκοσμιοποίηση για την υπόθεση από την Ελλάδα. Οδυσσίας Φωκάς. Ψηφίζουμε. Ηλεκτρονική ψηφορία. Πέρας. 43-5 εγκρίνεται. Πάμε στο επόμενο. Air France. Ψηφίζουμε. Πέρας. 40 υπέρ 5 κατά. Εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην τήση έκθεση Ευρωπαϊκής Τράπεζας για το 2013. Το τροπολογίες και 7 συγκριστικές. Κύριε Μαρτά, θέλετε το λόγο. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάτι, κάτι πάρα πολύ ε, σύντομο. Ο κύριος Κάζα ε, δημοκρατικά και ευγενικά ε, συμφώνησε με τις συμβατικές τροπολογίες Α και Γ, Α και Σ. Προσχωρήσαμε και εμείς αυτές και έτσι θα τις επιψηφίσουμε και με μεγάλη μας χαρά. Επομένως συμμετέχουμε σε αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες. Σας το λέω για να καταγραφεί στα πρακτικά της συνεδρίασης. Yes, we'll have that in the minutes. Σύμφωνοι. Καταγράφεται στα πρακτικά, λέει ο Πρόεδρος. Ψηφίζουμε τώρα. Συμβαστική Α, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Β. Κύριε Λένερτ Γι' αυτό που είπατε προηγουμένως, στη δική μου λίστα ψηφοφορίας δεν ε, αναφέρει το όνομά μου για την συμβαστική τροπολογία. Παρακαλώ να καταγραφεί και αυτό. Ναι, είναι και το δικό σου όνομα. Θα αναγραφεί. Το ίδιο επομένω και για τους σοσιαλδημοκράτες. Τρεις τέτοιες προσθήκες στα πρακτικά. Πάμε μετά στην παράγραφο Διορθώνει πρώτα τροπολογία 15. Υπέρ κατά και αποχές και εγκρίνεται. Check. Έλεγχος. The vote is closed. Πέρας της ψηφορίας. Εγκρίνεται. 16. Υπέρ. Κατά. Άποχες. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 25. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Έλεγχος για την 27. Ψηφίζουμε. Πέρασε. 33-14 εγκρίνεται. 28. Υπέρ. Συγγνώμη, καταπίπτει. Η 29. Δεν θα την ψηφίσουμε και πάμε στο 30. Υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παραγράφος 3. Τροπολογία 33 έως και 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, ε, συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτωτα. But we can check on that one. Θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 40. Πέρας ψηφορίας. Απορρίπτωτα. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος ηλεκτρονικός για το 46. Ψηφίζουμε. Πέρας. 25, 24. That was 45, wasn't it? 46. to 47. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Ποιο είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Ποιο είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τώρα του 48. Κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 49. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. αποχε Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. αποχε Εγκρίνεται. 51. Υπέρ. Κατά. αποχε Εγκρίνεται. Έλεγχος. Πέρα ψηφορίας. Εγκρίνεται. 29-20. Πάμε στο 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κατόπιν έχουμε την συμβαστική D. Δέλτα. υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 63. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ ψήφισε. There is a substitute. Okay, now it's okay. Α, ήταν κάποιος αναπληρωτής. Ε, Πορύπτεται. Ε, 24-27 περίπτωτα. Παράγραφος 5, τροπολογία 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτωται. Συμβαστική τροπολογία ε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το 73. Πέρας. 31 in favor. It's... 19 εγκρίνεται 74 και 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. F. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συγγνώμη, εγκρίνεται, διορθώνει η πρόεδρος. 80. Υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές Απολύτως G. Συμβαστική. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 80. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ Και τώρα έχουμε, λέει πρόεδρος, την τελική ψηφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης υπέρ. Α, όχι, λέει πρόεδρος, πρέπει να γίνει ηλεκτρονική ψηφορία και ψηφίζουμε τώρα. Πέρασε. 39 επτά Και τώρα να καλωσορίσω θερμά όσους συμμετέχουν στο speed hearing για την Ευρωπαϊκή Νεολαία. Ε, μεταδίδεται και στο διαδίκτυο αυτή η ακρόαση. Μπορεί να μας ακούσουν ε, και οι πολίτες από τα σπίτια τους. Εάν ε, θέλετε να σχολιάσετε και στο διαδίκτυο και επίσης βλέπετε και το hashtag για, ε, για την εκδήλωση αυτή θα παρουσιάζονται όλα αυτά ε, και στο Twitter ενώ διεξάγεται η ακρόαση και απλώς μια σύντομη εισαγωγή από μένα. Κύριε Μπάντα, είστε από την Ισπανία. Κυρία Ντεκλέβα είστε από την Σλοβενία και Γιωχάννα Νίμαν από τη Φινλανδία. Οι τέσσερις αυτοί νεαροί εκπρόσωποι της Ευρώπης θα είναι ένα καθοριστικό ε, πάνελ για το speed hearing για αυτήν την ε, ακρόαση express Για αυτούς τους νέους Ευρωπαίους που συναντήσαμε πριν τις εκλογές την Άνοιξη και που θα συνεχίσουμε να τους βλέπουμε και τα ερχόμενα πέντε χρόνια ελπίζουμε. Γι' αυτό θέλαμε να ακούσουμε ξανά εσάς και αυτά που θέλετε να ακουστούν σήμερα. Uh, να δώσω πρώτα το λόγο στο Ρικάρντο Δύο λεπτά. Θα μας παρουσιάσετε κάτι συναρπαστικό. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ε, βάσει των συζητήσεων για το AI, προτείνω ένα πρόγραμμα ανάπτυξης για τους νέους, διότι όταν αντιμετωπίζουμε το θέμα της απασχόλησης πρέπει να σκεφτούμε και τις συνθήκες επικατών στην Ευρώπη, την κρίση. Έτσι δεν μπορούμε με μικρά και μικροπρεπή μέτρα να λύσουμε μεγάλα προβλήματα. Είναι σημαντικό το επενδυτικό πρόγραμμα για την ε, Ευρώπη. Οι εργοδότες δεν θα μπορούν να προσλάβουν εργαζομένους άσχετα με το πόσο είναι ευέλικτοι ή πόση βοήθεια προσφέρει το κράτος. Δεν θα υπάρξει λοιπόν λύση εάν δεν υπάρξει και ανάπτυξη. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα ανάπτυξης για την Ευρώπη. Οι επενδύσεις είναι πάνω από όλα απαραίτητε για να αναθερμανθεί η οικονομία. Το πρόγραμμα Marshall ε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έβαλε την Ευρώπη στην ε, τροχιά της ανάπτυξης και πάλι και της ανα, Και πάλι στην Ευρώπη χρειαζόμαστε μια ανάλογη συμφωνία. 2% του ΑΕΠ για το μίσο πώ οι νέες τεχνολογίες, οι υποδομές, η έρευνα και η ανάπτυξη με πρόσβαση σε πιστώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με μείωση των τιμών της ενέργειας, όλα αυτά μπορεί να επιτρέψουν να ενισχυθεί η βιομηχανία και όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι το Συμβούλιο για, την, ε, ε, για, τα, για τους επαγγελματικού κλάδους λέει ότι μέχρι το 2016 θα έχουμε 6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, μέχρι το 2020 θα έχουμε 6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και αύξηση του ΑΕΠ. Επίση, η μείωση των φόρων σε περιοχέ με υψηλή ανεργία για να προσελκυστούν επενδύσει και επιχειρήσει, είναι και άλλε ιδέε. Αυτά θα επιβαρύνουν βεβαίω τα κράτη αλλά θα επιταχύνουν την ανάπτυξη τη Ευρώπη. Οι άμεσες επενδύσει μειώνουν τα επιτόκια και με τη συμβολή τη Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζα, αυτά μπορούν να συμβούν. Όμω, ε, αν δεν γίνει κάτι, μπορεί να χρειαστούν 20 έως 30 χρόνια για την ανοικοδόμηση τη Ευρώπη και έτσι θα έχουμε χάσει μια γενιά. Ευχαριστούμε Σοφία Ριμπέιρου. Αντίδραση από βουλευτή. Ευχαριστώ Πρόεδρε να συγχαρώ τους νέους που είναι εδώ σήμερα για αυτήν την πρωτοβουλία. Χρειαζόμαστε πραγματικά νέους που να αναλαμβάνουν δράση και θα είναι πολύ σημαντική η δράση σας ως νέων για το τι θα κάνουν και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είναι σημαντικό να μπορούμε να φροντίσουμε και τις δικές σας ανάγκες ως την πρότασή σας. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα βρίσκω ότι είναι διασκεδαστικότατο και ζητώ συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο να μιλάτε για πρόγραμμα Marshall για την απασχόληση και την ανεργία. Πραγματικά είναι σαν να έχει γίνει ένας πόλεμος. Οπότε πρέπει ε, να σας ευχαρώ για τον όρο που βρήκατε. Τώρα για όσα μας προτείνατε. Ανάγκη να ασχοληθούμε με το τι προσόντα έχουν οι νέοι. Εδώ ακούσαμε τι γίνεται με τους νέους και τη μακροπρόθεσμη ενεργεία και είδαμε να υπάρχουν σοβαρές αποκλήσεις μεταξύ των κρατών βάση βάσει των στοιχείων που διαθέτουμε, αλλά και εντός της κάθε χώρας. Πώς πιστεύετε λοιπόν ότι μπορούμε να υπερβούμε αυτό το εμπόδιο. Επίσης, προασπιστήκατε το 2% χρήση του ΑΕΠ για την καταπολέμηση τη ενεργεία. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα να προτείνετε, κάποια παρότρινση, καινοτομία, νέε τεχνολογίε. Σε ποιο τομέα πιστεύετε ότι πρέπει να επικεντρωθεί αυτό το κεφάλαιο. Ευχαριστώ. Μπράντο Ο κύριος Μπενιφέη. Ευχαριστώ και εγώ ήθελα να σας ε, συγχαρώ για αυτήν την ε, παρουσία σας. Πριν υπάρξει ο βουλευτής και εγώ έχω συμμετάσχει σε τέτοια προγράμματα και ξέρω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να ανταλλάξετε και τις απόψεις με τους πολιτικούς ηθήνοντες και για μας είναι πολύ ευχάριστο. Να πω ότι συμφωνώ με την ιδέα σας επειδή την προτείνατε έτσι όπως την προτείνατε, αλλά και εγώ ε, ήμουν ε, βουλευτής που συμμετείχα στην Πρωτοβουλία για την Ευρώπη Και χρειάστηκε να συλλέξουμε υπογραφέ με Ευρωπαίου πολίτε για να προτείνουμε ακριβώ αυτό που λέτε κι εσεί, ένα νέο πρόγραμμα Marshall, ε, ε μια πρωτοβουλία για την ανάκαμψη τη Ευρώπη. Εδώ όμω ε, ερχόμαστε στο θέμα των δημοσιονομικών δυνατοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή το ερώτημα είναι πώ θα χρηματοδοτηθούν όλα αυτά που λέτε. Νομίζω πρέπει να μα απασχολήσει αυτό, διότι όπω είπαν οι συνάδελφοι, έχουμε μεγάλε αποκλήσει μεταξύ των κρατών μελών. Ε, προβλήματα συνοχής και συνεκτικότητας, οπότε Χρειαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε, να απαντήσουμε και αυτό το ερώτημα. Με τι πόρους πιστεύετε ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε τις ιδέες σας. Εγώ πιστεύω ότι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να βρεθούν λύσει, όχι τα επιμέρου κράτη-μέλη να αναλάβουν δράση. Πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Πιστεύετε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, να προχωρήσουμε με, τον, ε, με τη φορολόγηση των συναλλαγών, των χρηματοδοτικών συναλλαγών λόγω χάρη. Ρικάρντο, τώρα να απαντήσετε και μετά. Ε, ναι, νομίζω έχω ένα λεπτό. Πολλές αλλαγές θα πρέπει να γίνουν, αλλά θα πρέπει να ζυγίσουμε το κόστος της ε, ανεργίας για τους νέους, για το Φαν, λέει 503 εκατομμύρια ευρώ και επομένω θα πρέπει να βρούμε κάποια μέτρα για να φρενάρουμε αυτή την ενεργή. Επίση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την φόρα αποφυγή, τη φορολογική απάτη και να βρούμε και άλλου τύπου επενδύσεων, ώστε να δημιουργηθεί κάποιο πλούτο. Τώρα, όσον αφορά αυτέ τι προτάσει για το πού θα βρούμε, πού θα επενδύσουμε, ε, για κάθε χώρα είναι διαφορετικά. Θα πρέπει να κάνουν γίνουν αλλαγέ στο παραγωγικό μοντέλο, να επαναβιομηχανίσουμε την Ευρώπη και πάλι, ή θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει εκεί που χρειάζεται αυτή η πίστοση και να αλλάξει το παραγωγικό πρώτο παραγωγικό μοντέλο κάθε χώρας. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ρικάρντο, δεύτερη ιδέα. Πάλι θα σας το πω στα ισπανικά, η δεύτερη υπόθεση η οποία βγαίνει από τις συζητήσεις του Άγιος Δεβέντη είναι ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τις επενδύσεις στη νεολαία. Έχουμε αυτή την ε, ακραία λιτότητα που δεν βιαλτίζει τα πράγματα όσον αφορά την Τι να κάνει χειρότερη διατάση. Οπότε αυτό ιδίω αφορά την ποιότητα ζωής του Πολωνίου και θα πρέπει να εστιάσουμε τη ζήτησή μας στο πώς θα μειώσουμε τον εθνικό προπολογισμό και τον ε, ευρωπαϊκό πληθυσμό. Αντί για αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε στο μέλλον κάποιες ε, ε, επενδύσεις. Είχαμε περικοπές στην παιδεία, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και τελικά περισσότερα ευθύγησαν οι νέοι. Τελικά οι νέοι κινδυνεύουν περισσότερο από αυτή την κρίση από ότι οι ηλικιωμένοι. Επομένω, πρέπει να γίνουν τέτοιε επενδύσει, επενδύσει για την ζήτηση στην αγορά εργασία, αλλά επίση ε, τα μέτρα που έχουμε λάβει είναι ανεπαρκή, δεν εφαρμόζονται καλά και επομένω χρειάζονται 6 δι ε, ευρώ και όχι 21 όπως προτείνει η διεθνή Γραφείο εργασία, αλλά πέραν του οικονομικού και κοινωνικού κόστους της ε, της ανεργίας. Επομένως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ευρωπαϊκές συστάσεις, οπότε θα πρέπει να δείξουν τη γνώμη τους στον προγραμματισμό, την αξιολόγηση των προγραμμάτων και τη διαχείρισή τους είναι. Αλλά πρέπει να πάμε πάρα πέρα και θα πρέπει να διαλέξουμε το πώς θα έχουμε ενεργητικές, δυναμικές, πολιτικές επασχόλησης, κοινωνική πρόνοια υπέρ της νεολαίας, να βοηθήσουμε αυτούς που χρειάζονται περισσότερο. Να έχουμε επίσης κάποιο είδους συνέπεια και συνοχή ε, για την ε, για την νεολαία. Να σταματήσουμε τις περικοπές που σταμάτανε τη ζήτηση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Να προσέξουμε την παιδεία, την ποιότητα των μήλων, τη ζωή, ζωής, των νέων και επομένω θα πρέπει να υπάρχουν κάποια προγράμματα μακρόπνοα. Να γίνει καινούριο δημοσιονομικό προγραμματισμό, αυτό που να χαρακτηρίζεται από αλληλεγγύη, να είναι προοδευτικό, να καταπολεμήσουμε την κοινωνική, ε, την τον κοινωνικό αποκλεισμό αυτών των πλέον. Ε, Ευχαριστώ, Γιωχάννα. Η δεύτερη ιδέα σου τώρα. Επαναρχόμαστε στο ζήτημα που τέθηκε νωρίτερα για τις πρακτικές ε, ασκήσεις. Είναι πολύ σύνηθες ε, μεταξύ των νέων να κάνουν πρακτική άσκηση. 50% των νέων έχουν κάνει ιδιαίτερα σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς όσον αφορά την απασχόληση και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Οι πρακτικές ασκήσεις μπορούν πραγματικά να αποτελέσουν τη, γέφυρα για τη μετάβαση στην αγορά εργασίας, αλλά υπάρχουν προβλήματα. Μόνο 40% των ε, ε, ασκούμενων αμείβονται 30% δεν έχουν συμβόλαια, 30% επίσης έχουν χαμηλής ποιότητας πρακτικές ασκήσεις και κακές συνθήκες εργασίας στο χώρο εργασίας τους. Το ερώτημα είναι, έχει ο καθένας την οικονομική δυνατότητα να κάνει πρακτική άσκηση. Μήπως η απλήρωτη εργασία αντικαθιστά την πληρωμένη εργασία και μήπως αυτό οδηγεί τους ανθρώπους να μην έχουν δυνατότητα να μαθαίνουν και να αποκτούν θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας. Η συγκεκριμένη μας ε, σύσταση, πρόταση, είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπερασπιστεί τη φωνή των νέων ανθρώπων σε τρεις τομείς. Πρώτον, να υπάρχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο για, ε, στην πρακτική άσκηση. Δεν δουλεύουμε τζάμπα, αλλά για κάποιο λόγο. Δεύτερον, αμοιβή για τους ε, ασκούμενους. Και τρίτον, όπως είπα, το θέμα μας δεν είναι να υποκαθιστούμε την πληρωμένη εργασία, αλλά να αποκτάς και κάτι και στο τέλος ε, και η στόχοι μιας πρακτικής άσκησης θα πρέπει να είναι σαφείς σε όλους όσους εμπλέκονται. Εμείς θέλουμε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου ε, σε όλα αυτά τα ζητήματα. Υπήρξε ε, και μία κίνηση από το Συμβούλιο, αλλά δεν, δεν αναφέρθηκε το Συμβούλιο σε, αυτά τα, σε αυτούς τους τρεις άξονες που αναφέρθηκα. Θέλουμε η εθνική νομοθεσία να ορίζει τι ακριβώς περιλαμβάνει μια πρακτική άσκηση και τι ακριβώς συνιστά ποιοτική πρακτική άσκηση. Υπάρχει επίσης η χάρτα τον, ε, για, τις, για την πρακτική άσκηση που περιγράφει όλα αυτά τα στοιχεία που ανέφερα. Η Χέλκα Στίβενς Ευχαριστώ. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το οποίο είπαν οι φιλοξενούμενοι μα νέοι όσον αφορά τα η stage. Πολύ ενδιαφέρον για όσους ε, συμμετέχουν ακριβώς πώς πληρώνονται κλπ. λοιπά. Επίσης και για το σκοπό το τελικό θα πρέπει να δούμε τι γίνεται, τι θα πρέπει να μάθει κανείς στην πρακτική και αυτό είναι το πλεονέκτημα για τους ε, νέους, το βασικό πλεονέκτημα. Πάντοτε πρέπει κανείς να παρακολουθεί τι γίνεται. είναι ζητούν έργο, δουλεύουν και κατόπιν θα πρέπει φυσικά να αμυφθούν από τον εργοδότη και βέβαια πάσα συνθήκη θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο οπότε θα πρέπει βέβαια να είναι κανείς πάρα πολύ προσεκτικός διότι υπάρχουν επιπτώσεις από αυτά όσον αφορά την εμπειρία, την επαγγελματική που θα αποκτήσουν οι νέοι. Ακριβώς υπάρχει και αυτή η πτυχή που ισχύει με την κατάρτιση και θα πρέπει επομένω και επίσημοι φορείς να σκεφτούν τι σχέση έχει περίοδος μαθητείας με την πραγματική δουλειά, τι κάνει δηλαδή στην πράξη. Συμφωνούμε απολύτως. Ότι γίνεται σε πάρα πολύ επικίνδυνες συνθήκες ε, ε, αυτός ο θεσμός των ε, στάζ. Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη να είναι όλα ασφαλή για 100% και θα πρέπει αυτό κάπου να αναγραφεί. Αυτό, είναι ο σκοπός που θέλουμε. Τάνια. Hola, muchas gracias. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό το οποίο βλέπουν είναι τι κίνδυνος υπάρχει, πόσο ευάλωτες είναι οι θέσεις απασχόλησης. Πάμε για περίπου 50% στην Νότια Ευρώπη για την ενέργεια των νέων. Όμως αυτές οι υποτροφίες, αυτές οι μαθητείες δεν κάνουν τίποτα. Ουσιαστικά εξασφαλίζουν ε, δωρεάν ή φτωχές ε, θέσεις απασχόλησης. Αποκλείται πάρα πολύ νέοι γίνονται τελικά εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα. Επομένως, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να αναφέρουμε κάποια παραδείγματα. Ποια είναι τα δικαιώματα, ποια είναι τα όρια στα οποία μπορεί να φτάσει κανείς κατά την, ε, ε, κατά, κατά την περίοδο εκμάθησης και με τις συμφωνίες της πανεπιστημιακές και όσον αφορά τις επιχείρησεις. Πάντοτε υπάρχει κάποια υποτροφία που έχει αποζημίωση. Δεν θα πρέπει ε, το αντίθετο να γίνεται βάρος. Και θα ήθελα να ρωτήσω τη Γιωχάννα. Δεν έχουμε χρόνο να το πούμε σε βάθος, αλλά αυτοί που πέρασαν από γη, τι εμπειρία έχουν. Πώς είναι δυνατόν να μην καταλήξουμε μια υποτροφία σε μια τέτοια ε, μαθητεία με τέτοια συνέπειες, αλλά να καταλήξουμε σε κάποια πραγματική θέση απασχόλησης ναι, η πρακτική άσκηση πρέπει να ωφελεί τον νέο και οι δυνατότητε πρακτική άσκηση είναι διαφορετικέ για διαφορετικού άνθρωπους. Για παράδειγμα, στο πανεπιστήμιο είναι διαφορετικό το να παίρνει κρατική ενίσχυση, χρηματοδότηση. Ίσως τότε θα μπορούσε να το συζητήσουμε το ζήτημα, αν θα αμείβεσαι ή όχι. Αλλά στην ανοιχτή, στην ε, ιδιωτική αγορά, ε, φυσικά αν πηγαίνει και κάνει πρακτική άσκηση θα πρέπει να, να αμείβεσαι. Κανείς δεν μπορεί να ζήσει με αέρα κορπανιστό και είναι πρόβλημα αυτό για μας. Επίσης ε, το ζήτημα της αποζημίωσης για τη μετακίνηση στο χώρο εργασίας, τέτοια θέματα είναι ζητήματα όπου θα πρέπει να υπάρχει νομοθεσία που θα ορίζει τι αποτελεί υψηλής ποιότητας πρακτική άσκηση και τι όχι. Και πρέπει να δημιουργήσουμε κοινά πρότυπα, διότι χωρίς αυτά μπορεί ο καθένας να δημιουργήσει πρακτικές ασκήσεις με βάση τις δικές του ε, επιθυμίες. Και αυτή τη στιγμή η πρακτική άσκηση τίνει να γίνει τζάμπα εργασία για τις επιχειρήσεις και αυτό είναι απαράδεκτο. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην πέμπτη από τον Τζόναθαν Μακ. Thank you Ευχαριστώ πολύ. Θα επικεντρωθώ στην διεθνή διακρατική κινητικότητα των νέων. Βάσει των ιδεών που αναφέρθηκαν και στην εκδηλωσία στο Στρασβούργο, πρότεινα στα μέλη του ε, Κοινοβουλίου να προβλέψουν προγράμματα και μέτρα ώστε να έχουν ίσες ευκαιρίες και συμμετοχή ε, οι νέοι στα προγράμματα κινητικότητας. τα προγράμματα διεθνούς κινητικότητας, όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντών, είναι μια τεράστια ευκαιρία για τους νέους, για να αναπτύξουν τις διαπολιτισμικές τους δυνατότητες, τις γλωσσικές τους δεξιότητες και την ευκαιρία να πετύχουν ως νέοι ενήλικοι στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, θεωρούμε και το αποδεικνύουν και πολλές μελέτες ότι αυτά τα προβλήματα κινητικότητας εμποδίζουν ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, ιδίως τους νέους με τα ανώτατα εκπαιδευτικά προσόντα. Η πρόσβαση στην κινητικότητα είναι πολύ σπάνια και δύσκολη για τους ανθρώπους από δύσκολες ομάδες του πληθυσμού όπως τους Ρωμά ή άλλες εθνοτικές μειονότητες. Η έλλειψη γλωσσικών δεξιοτήτων είναι ένα κριτήριο αποκλεισμού για πολλούς νέους ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στα προγράμματα εθελοντών και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Επισήμω όμω αυτά τα κριτήρια δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και να εφαρμόζονται. Προτείνω λοιπόν στο Κοινοβούλιο να ασκήσει πολιτική πίεση ώστε να υπάρχουν ίσε ευκαιρίε και να υπάρξει ένα ποιητικό αντίκτυπο στην ίση μεταχείριση όλων στα προγράμματα αυτά κινητικότητα. Μέσω τη γλωσσική εκμάθηση και τη προσφορά δεξιοτήτων στου νέου θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η βελτίωση των ίσων ευκαιριών για να υπάρχει αποτελεσματικότητα, ποιότητα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα ότι μπορούν να πετύχουν τα προγράμματα κινητικότητας. Γι' αυτό χρειάζονται και μηχανισμοί παρακολούθηση και αξιολόγηση που είναι αυστηροί και να παρακολουθούν τη συμμετοχή των Ρωμά, των μεταναστών και των νέων από μειονοτικέ ομάδε του πληθυσμού. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ, Τζόναθαν Μακ, για τις ιδέες σου. Μπορώ να τις στηρίξω, αλλά είναι σημαντικό και εγώ πιστεύω η κινητικότητα να αυξηθεί γενικότερα στην Ευρώπη. Πόσο μάλλον ε, στα προγράμματα που ήδη έχουμε στην Ευρώπη. Επίσης πιστεύω ότι σημαντικό είναι να κοιτάξουμε τις ε, συνθήκες που ισχύουν στις διαφορετικές χώρες. Πώς δηλαδή μπορεί κανείς να καλύψει όχι μόνο την γενετικότητα αλλά λόγω χάρη και την πτυχή της ασφάλειας. Ξέρετε, είμαι από την Δανία και συχνά μιλάμε για την ελαστασφάλεια, ε, την ασφάλεια με ευελιξία. Είναι ε, αυτή η δυνατότητα δημιουργίας ε, ευελιξία, περισσότερης ευελιξίας, αλλά πρέπει να δούμε και τη διάσταση της ασφαλούς εργασίας, της βεβαιότητας. Ευχαριστούμε κύριο Φουντούλη. Αγαπητέ Τζόναθαν, σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα εδώ και μοιράζεσαι μαζί μας την ιδέα σου σχετικά με την κινητικότητα των νέων στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ένα πρόγραμμα ίσων ευκαιριών για την νεολαία προσφέρει στους συμμετέχοντες, δηλαδή σε εσά τους νέους, μεγάλα ωφέλη. Μήπως όμως αυτό που εσύ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ονομάζετε κινητικότητα ερμηνεύεται ως δημιουργία σύγχρονων μορφών εργασιακής εκμετάλλευσης. Οι περισσότερες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται είναι προσωρινές και χαμηλά αμοιβόμενες. Εκτός από τον κίνδυνο της καταπάτησης από κάποιους κάθε εργασιακού δικαιώματος, μοιραία κινητικότητα οδηγεί και στην ουσιαστική ερήμωση των χωρών που αυτή τη στιγμή έχουν χειρότερες εργασιακές συνθήκες από κάποιες άλλες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, από τη στιγμή που θα στερήσουμε από χώρες όπως τη δική μου, την Ελλάδα, το σημαντικότερο παράγοντα για μια μελλοντική ανάπτυξη, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, τους νέους και τα καλύτερα μυαλά της χώρας, πώς μπορούμε να περιμένουμε ένα καλύτερο μέλλον. Σκέφτηκες ότι αυτό το εκμεταλλεύονται οι πιο ισχυρές χώρες. Δηλαδή την εκμετάλλευση των ταλαντούχων νέων των πιο αδύναμων οικονομικά κρατών για δικό σου όφελο. Επιπλέον, η πρότασή σου για την Ευρώπη του μέλλοντο είναι η δημιουργία εργαζόμενων δύο ταχυτήτων, αυτών που θα έχουν τη δυνατότητα να μεταναστεύσουν αναζητώντα ένα καλύτερο αύριο και των ανεδίκευτων που θα μείνουν πίσω σε μια ηρεμωμένη χώρα. Σε ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ, η απάντησή σου. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πιστεύω και είμαι πεπισμένος ότι τα προγράμματα κινητικότητας έχουν ε, την αξία τους. Θα πρέπει βεβαίως να δούμε και τις συνθήκες ε, που θα εξασφαλίζουν αυτή την ποιότητα, όπως και την σταθερότητα. Ε, οι νέοι θα πρέπει να κάνουν τις επιλογές τους ως αυτόνομα άτομα, ανεξάρτητα άτομα. Για από αυτήν την οπτική γωνία πρέπει να τονίσω ότι θα πρέπει να προσέξουμε η κινητικότητα να μην γίνει ένα όχημα ώστε η ανώτατη μεσαία τάξη ε, να ε, επωφεληθεί μόνο εκείνη, αλλά και οι νέοι με λιγότερες ευκαιρίες, με λιγότερες δυνατότητες. Ιδίως ε, οι νέοι με ιστορικό και με προέλευση που δεν τους έχει δώσει πολλά εφόδια θα πρέπει να αποφύγουν τις καταστάσεις αποκλεισμού. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Και τώρα μπορείτε να περάσετε στη δεύτερη ιδέα σας. Πάρα που έχουν συμμετέχει σε αυτό το ΑΕΛ, λένε ότι ανησυχούν πάρα πολύ όσον αφορά την ακραία δεξιά, όσον αφορά την ξενοφοβία και τον ρατσισμό στην Ευρώπη. Και εν ώψη των ευρωεκλογών τότε είχαμε πει πολλοί από εμά ότι δεν υπάρχει χώρο για τέτοιου είδου ακροδεξιά κόμματα και ακροδεξιέ ιδεολογίε στην Ευρώπη. Στο Στασβούργο δεν είχαμε πει ότι εκατοντάδε χιλιάδε από Ρωμά, ανηλίκου και ανηλίκου, υφίστανται δεσμενεί διακρίσει, ε, apartheid στο σχολείο, κοινωνικό αποκλεισμό και πάρα πολλές ε, ε, πολιτικές για την κοινωνική συμπερίληψη ε, και κοινωνική ένταξη στοχεύουν στους Ρωμά που φέρνουν από γενοκτονίες, από διώξεις και πάρα πολλοί θεωρούν ότι είναι οι στόχοι της καταστολής η Ρώμα. Δεν θα γίνει τίποτα αν δεν υπάρξει κάποιο είδου δράση από τα κοινοβούλια και να κάνουμε κάτι για τους Ρωμά και για την, ε, τους νέους τσιγκάνους. Οπότε θα πρέπει η κοινωνία να αναγνωρίσει τον ιστορικό τους ρόλο και επίσης την θέση τους. Ε, οπότε θα πρέπει να υπάρξει κάποιο είδου συμφιλία, κάποιο αναγνώριση. Και όλοι είναι ε, στο ΑΕ και η Ρώμα και η μη Ρωμά είπαν ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί η γενοκτονία στον Ρωμά που είχαμε 500.000 στον Ρωμά οι σκοτώθηκαν από τους Ναζί στην Ευρώπη. Το 2014 είναι η 70η ε, επέτειος 7ης Αυγούστου που είχαμε αυτή τη γενοκτονία και είχαμε πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναγνωρίσει την γεροκτονία κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ότι θα πρέπει να ανακηρυχθεί η Δευτέρα Αυγούστου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας. Σας προτείνω να γίνει μια τέτοια πολιτική που να συνοδευτεί από ένα πρόγραμμα ε, κατά του ολοκαυτώματος και υπέρ της ε, εκπαίδευσης και να γίνει αυτό επίσης μια ε, προτεραιότητα σε διάφορα προγράμματα, ιδίως δε του προγράμματος Erasmus. Moi, je voudrais euh, euh, déjà vous, vous remercier. Ήθελα να σας ευχαριστήσω και είναι μεγάλη μου χαρά που σας ξαναβλέπω εδώ στις Βρυξέλλες αφού σας συνείδησα πρώτη φορά στο Στρασβούργο τον ε, Μάιο. Ε, για όσα αναφέρατε για το θέμα των Ρωμά που κατά τη δική μου την άποψη έχει να κάνει ούτως ή άλλως με κάθε μορφή διακριτικής μεταχείρισης. Πιστεύω όλοι θα συμφωνήσουμε ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τις μορφές διακριτικής ε, μεταχείρισης, όποιες και αν είναι αυτές όλο το Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και μιλήσαμε και χθε ε, γι' αυτό, για τι ε, διακριτικέ μεταχειρήσει γενικότερα, για ορισμένε ομάδε του πληθυσμού όπω η Ρωμά ή τα άτομα με αναπηρίε και ούτω καθεξής. Αναφέρατε το θέμα του Εράσμους ΣΥΝ. Είμαι πολύ ε, ευνοϊκή σε αυτό που είπατε και σε γενικέ γραμμέ νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε για του νέου. για να τονώσουμε την επιχειρηματικότητα, να καταπολεμήσουμε τις ε, μορφέ διακριτική συμπεριφορά. γενικότερα να στηρίξουμε όλο τον πληθυσμό, χρειαζόμαστε στήριξη ε, σε τοπικό επίπεδο. Οι νέοι δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφορία πολλέ φορέ, είτε για τα δικαιώματά του, είτε για τα διάφορα προγράμματα που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, για αυτόν τον λόγο θα πρέπει την πρόσβαση να την εξασφαλίζουν οι αρχές τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να μπορούν να αναδεικνύουν τα διάφορα προγράμματα. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπαλά. Ναι, το πρόβλημα σήμερα είναι ότι όντως έχουμε δύο νεολαίες. Ε, την νεολαία που παρά την κρίση καταφέρνει να αναλάβει ενεργό ρόλο και μια άλλη που αισθάνεται την απόρριψη όλο και περισσότερο και έχει γνωρίσει τις σοβαρότερες συνέπειες από την ε, εγκατάλειψη του σχολείου ή από τις διακριτικές μεταχειρήσεις, τις μορφές διακριτικής συμπεριφοράς. Για τους Ρωμά, τους νέους Ρωμά ισχύει αυτό και πολλές φορές προσπαθούν να ξεφύγουν από το πεπρωμένο τους, πολλές φορές προσπαθούν να ξεφύγουν από την ίδια την οικογένειά τους ε, για να ζήσουν διαφορετικά στις ε, περιοχές τους. Όμως πολλές φορές πέφτουν θύματα δικτύων που έχουν δυστυχώς παράνομες και απαράδεκτες ε, δράσεις. Όχι πάντα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε πρώτα την ιστορία τους, την πορεία τους, πριν τους εντάξουμε στις κοινωνίες μας. Δεν θέλουμε να έχουμε ένα πολιτιστικό διαχωρισμό αναγνωρίζοντας μια ταυτότητα που είναι μια ταυτότητα ε, αρνητική, αλλά να παραδεχτούμε ότι οι Ρωμά αποτελούν μέρος της ιστορίας της Ευρώπης εδώ και αιώνες. Οπότε το να ε, βλέπουμε σήμερα ότι μεγάλα δράματα ή μεγάλες ε, σελίδες της ιστορίας μας έχουν γραφτεί με τη συμμετοχή των Ρωμά, όπως αυτό που αναφέρατε εσείς για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι συνέβαλαν στην διαμόρφωση του πολιτισμού μας, είναι σημαντικό. Πρέπει να το πούμε μια και καλή. Οι νέοι Ρωμά και οι Ρωμά ε, σε κάθε περίπτωση είναι Ευρωπαίοι με πλήρη δικαιώματα και μπορούν να συμμετάχουν στο κοινό μας προμένο για να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε. Γιώναταν, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Το να αναγνωρίσει κανείς ε, τις επιπτώσεις των διακριτικών μεταχειρήσεων στην ζωή των Ρωμά είναι σημαντικό. Πολλοί άνθρωποι από τους Ρωμά νιώθουν ότι έχουν τόσο ισχυρό στίγμα που φοβούνται να ε, ζήσουν τη ζωή τους με βάση την ταυτότητά τους. Και το καλοκαίρι στην Κρακοβία και στο Auschwitz έγινε συνάντηση πάνω από χιλίων ε, Ρωμά και διαπιστώσαμε ότι πρέπει να γίνει αναγνώριση ε, αιώνων ιστορίας και αυτό χρειάζεται πολιτική ε, αναγνώριση. Η Γερμανία αναγνώρισε την γενοκτονία των Ρωμά μόλις το 1982 στο παρελθόν υπήρξε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά μέχρι στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει αναγνωρίσει την γενοκτονία κατά τον Ρωμά και ελπίζω αυτό να γίνει πολύ σύντομα. Ε, ευχαριστώ πολύ. Κάγια Ντέκλεβα. Θα μας παρουσιάσεις την έβδομη ιδέα, τη δική σου ιδέα. Ευχαριστώ πολύ. Το πρώτο θέμα για το οποίο θέλω να μιλήσω είναι η υψηλή ποιότητα θέση εργασία για νέους. Για να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής ζωής και η εργασία των νέων πρέπει να δημιουργηθούν υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας για τους νέους. Ο, ε, η Διεθνή Οργάνωση Εργασίας προβλέπει ότι η νεανική ανεργία θα συνεχίσει να είναι πρόβλημα για τα, τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια. Έτσι, πολλοί νέοι βρίσκονται σε ένα φαύλο κύκλο οι νέοι άνθρωποι ως δημογραφική ομάδα έχουν διαφορετικές ανάγκες, αξίες και διαφορετικές γνώσεις και όλα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την πρόσληψη ενός νέου ανθρώπου. Οι χαμηλή ποιότητα θέσει εργασία που δεν λαμβάνουν υπόψη τι διαφορέ των νέων δεν είναι καλέ. Εκτό από το ότι είναι σταθείς μπορεί να, έχουν, να οδηγήσουν σε πολύ σοβαρέ επιπτώσει, για παράδειγμα κατάθλιψη. Οι νέοι άνθρωποι αξίζουν να έχουν καλύτερες ε, ε, θέσεις απασχόλησης, ε, όχι υποαμοιβόμενε και κακών συνθήκων. Οι νέοι άνθρωποι βρίσκονται σε πολύ ευάλωτη φάση τη ζωή τους. Αυτό που θέλω να προτείνω είναι μια, μια νέα πράξη νομοθετική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να αφορά τους εργοδότες και να θεσπίζει συγκεκριμένα πρότυπα εργασίας που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητας των νέων ανθρώπων. Αυτό θα συνοδεύεται από μια εκστρατεία για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τους νέους που εργάζονται σε χαμηλής ποιότητα θέση εργασία. Επίση, για την, οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν τους εργοδότες τους και να τους δίνουν συμβουλέ για το πώ θα μπορούσαν να καθοδηγήσουν και να βελτιώσουν τον χώρο εργασία τους. Οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει να θεωρούνται ω πηγή συνεισφορά στην κοινωνία και όχι ω βάρο για την κοινωνία. Ευχαριστώ, ο Άνταμ Κώσα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι βρίσκω εξόχως ενδιαφέρουσα τη συζήτηση σήμερα, διότι γίνεται συζήτηση για πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Η Επιτροπή μας ασχολείται εδώ και χρόνια με τα θέματα αυτά. Οπότε πραγματικά βρίσκεστε στο, καταλληλότερο σημείο για να κάνετε αυτή τη συζήτηση. Έχουμε πολλές φορές απασχοληθεί, ασχοληθεί με τις θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και πολύ συχνά ανακύπτει το ερώτημα πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ε, εκπαιδευτικά συστήματα υψηλής ποιότητας, πώς θα μπορούν όλα αυτά να ενταχθούν και στην ανώτερη εκπαίδευση, ώστε να μπορούν να έχουν και αντίκτυπο στην αγορά εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι οι θέσει απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 35% είναι θέσεις απασχόλησης που ε, απαιτούν υψηλές δεξιότητες και γι' αυτόν τον λόγο οι νέοι άνθρωποι οφείλουν να έχουν λάβει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στο μέλλον η τεχνολογία πληροφορικής θα εξελιχθεί ακόμη περισσότερο και αυτό θα οδηγήσει σε κατάργηση πολλών θέσεων εργασίας. Βεβαίως θα δημιουργήσει και κάποιες νέες θέσεις εργασίας, αλλά θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, σε ποιο βαθμό δηλαδή η τεχνολογία πληροφορικής θα δημιουργήσει ή αντίστοιχα θα καταργήσει θέσεις απασχόλησης και αν και κατά πόσο οι εργοδότες είναι σε θέση να προσαρμοστούν στις ανάγκες αυτές. Η ε, κυρία Χάρκιν, ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστούμε. Είναι πολύ σημαντικό κάποιο να έρχεται και να προτείνει μια λύση, όχι μόνο να μιλάμε για τη διάσταση των προβλημάτων, γιατί τα προβλήματα τα γνωρίζουμε καλά. Όντω, η πιο πρόσφατη έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η τριμηνία έκθεση για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην Ευρώπη, ε, εντοπίζει ότι για όλου κάτω των 25, 40% που είναι ε, στον ενεργό πληθυσμό είναι ως επιτοπλίστων κατά τα δύο τρίτα με προσωρινά συμβόλαια, προσωρινές συμβάσεις ή σε ε, εργασία μερικού χρόνου. Αυτό δείχνει τι τάση υπάρχει και γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε κάποια λύση. Μιλήσατε για την ε, αύξηση τη φτώχεια. Σήμερα το πρωί στη συζήτησή μα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλούσαμε για περισσότερου, 8 εκατομμύρια περισσότερου φτωχού το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, άκουσα αυτά που είπατε και εσείς και η Γιωχάνα για ποιότητας πρακτικές ασκήσεις και ποιότητας θέσει εργασίας. Βλέπω την ανάγκη να υπάρξουν κάποιοι στόχοι, αλλά θα θέλατε να είναι δεσμευτικοί, να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο σε συνδυασμό με κάποια χάρτα ίσως για τις πρακτικές ασκήσεις, για τα stage, για να ε, προσπαθήσουμε να καλέσουμε τα κρατημέλη, να δουν τις βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν ε, ανά την Ευρώπη και να ανταλλάξουν γενικώ πληροφορίες. Γίνεται πολύ πολλής λόγος για την βελτίωση των δεξιοτήτων, την αλλαγή επαγγελματικού προσανατολισμού, για την ε, εκ νέου κατάρτιση. Πολλοί όμω είναι οι νέοι που όλο αυτό το στάδιο το έχουν περάσει και είναι έτοιμοι να εργαστούν. Εκεί είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να ε, καταλάβουμε καλά. Διαφορετικέ ανάγκε και διαφορετικέ γνώσει. Αυτό είναι συνήθω το πρόβλημα και θα πρέπει να ε, κάνουν κάτι γι' αυτό και οι εργοδότε από την πλευρά του. Κάγια, η αντίδρασή σα. Ευχαριστώ σε ό,τι αφορά την πρώτη σας ερώτηση, να ξεκινήσω λέγοντας ότι η πληροφορική και δημιουργεί αλλά και αφαιρεί θέσεις εργασίας. Παρόλα αυτά υπάρχει ε, ανάγκη για κάποιες βασικές θέσεις σε τομείς όπως ο κατασκευαστικός, στα σφαγεία και ούτω καθεξής. Ε, βεβαίως, οι νέοι μερικές φορές δεν θέλουν τέτοιες δουλειές. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα, μια κατάσταση λίγο διφορούμενη. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε όχι μόνο τις θέσεις που προσφέρονται χάρη στις τεχνολογικές λύσεις και τις νέες τεχνολογίες. Ε, επίσης, για τη δεύτερη παρατηρήσή σας, όπως και εσείς είπατε αυτά, ίσως θα μπορούσαν να διασυνδεθούν με την χάρτα των ε, ε, πρακτικών ασκήσεων ποιότητας εφόσον δημιουργηθεί. Αλλά αυτά πρέπει να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα σημαντικό μας συνομιλητής εδώ είναι ακριβώς το φόρουμ της Ευρωπαϊκής Νεολαίας. Με την διάρθρωση της ε, οργανώσης νεολαίας, και εμπειρογνωμόνων. Εκεί μπορούμε να έχουμε μια σημαντική συμβολή. Πρόεδρος, ευχαριστούμε και τώρα μπορείς να μας παρουσιάσεις τη δεύτερη ιδέα σου. Η δεύτερη μου ιδέα παραμοιασμένη πρώτη αφορά τη δημιουργία ε, σχέσεων, διάβλων μεταξύ ε, της μαθίας και της ε, αγοράς εργασίας να δούμε πώς γίνεται να τον έχουμε τόσο πολλούς που δεν έχουν δουλειά και είναι τελικά θέμα της αγοράς εργασίας. Μπορεί να λυθεί το πρόβλημα, μπορεί αυτό να γίνει με περισσότερη συνεργασία αυτών των δύο τομέων, οπότε θα πρέπει ο καθένας να αποφασίζει για το μέλλον του στην παιδεία. Ε, όμως χρειάζεται πληροφορίες με τις προοπτικές, της αγορά εργασίας και τις δυνατότητες στο μέλλον. Και μία από τις λύσεις, κατά ναι, είναι να προσέξουμε το εκδοτικό σύστημα, να συνδυάζει τη θεωρία με την ε, πρακτική και την πράξη, οπότε ό,τι μαθαίνουμε στο σχολείο μετά να ισχύει για την περίοδο μαθητείας, οπότε και έτσι ε, σχετίζονται ε, με τους εργοδότες και με την αγορά εργασία. Έχουν εμπειρία οι νέοι, έχουν ό,τι χρειάζεται ούτως ώστε να αποφασίσουν σωστά για το μέλλον τους. Και έτσι έχουν ό,τι χρειάζεται για τον ανταγωνισμό. Πάρα πολύ καλό αυτό. Και για τους εργοδότες και για τους νέους. Ο ένας μαθαίνει από τον άλλο. Ένα καλύτερο επιδοτικό σύστημα σημαίνει σύνδεσή του με την αγορά Εργασία, συστημική ενέργεια, αποτελεσματική και μακρόπνοη. Σαν την εγγύηση για τους νέους να ισχύει για όλη την Ένωση. Και είναι θέμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να φροντίσει τους νέους, να τους εξασφαλίσει μέλλον. Θυμάστε, στην προηγούμενη εκστρατεία τα είχατε πει αυτά, ήρθε η ώρα των έργων. Yeah, thanks. Before I start, I also wanted to say... Αν και πρώτα πρώτα να σας πω ότι με μεγάλη μου χαρά βλέπουμε επιτέλους εδώ να έρχονται και κάποιοι νέοι. Δεν είναι αυτό καθημερινό φαινόμενο. Σας ευχαριστούμε και πάλι για όσα είπατε και μία από τις ιδέες που μας δώσατε είναι αυτός ο, ο του Twitter και τώρα είμαστε δραστήριοι και ε, στα ψηφιακά. Να μια ιδέα που μας δώσατε. Οπότε τώρα για να δούμε κάτι σε σχέση με αυτά που μας είπατε. Υπάρχει αυτό το, το, το, το στο μεταξύ δεξιοτήτων και ε, δουλειάς. Και επομένως ε, θα πρέπει να γίνει την παιδεία και έτσι να έχει πιο πρακτικό χαρακτήρα. Πρέπει να είναι πιο προσανατολισμένη η παιδεία και η εκπαίδευση. Να μπορούν οι νέοι να έχουν κατάλληλη παιδεία. Αυτό βέβαια από τη μακρόπνο σχεδιασμό. Και βέβαια υπάρχουν τις ανεργίες, οπότε αυτό είναι άλλο θέμα. Τέλο πάντων, θα πρέπει να υπάρξει και κάποιο πρόγραμμα και κάποιε ιδέε ε, πρόθεσμο χαρακτήρα. Και, όπω είπατε, να ισχύουν όλα αυτά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τα παιδιά πρώτα απ' όλα γιατί είναι τόσο ωραίο να βλέπουμε νέους που να έρχονται εδώ στο κοινοβούλιο και να μας προτείνουν συγκεκριμένα πράγματα για την αλλαγή. Αυτό είναι κίνητο για το Ευρωπαϊκό Γενοβούλιο και τη θεσμικά όργανα τόσο ώστε να ξεκινήσει καινούργιε ε, δράσει. Γιατί πάρα πολύ συχνά λέμε ωραία πράγματα, αλλά χρειάζονται συγκεκριμένε δράσει. Ε, να, γιατί χρειάζεται το κίνητρο. Οπότε όσον αφορά αυτό το είδος την διασύνδεση, την καλύτερη διασύνδεση μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και του κόσμου της δουλειάς. Συμφωνώ 100%. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να έχουμε λιγότερη θεωρία και περισσότερη πρακτική κατά την περίοδο εκπαίδευση και μαθητείας των νέων. Και σε αυτό το σημείο το πανεπιστημιακό ιταλικό σύστημα ε, δεν προσφέρει πάρα πολύ γιατί έχει πολλή θεωρία και λίγη πρακτική. Άρα θα πρέπει να βάλουμε περισσότερα από τον πραγματικό κόσμο της, της στα πανεπιστήμια και αυτό θα βοηθήσει και τους νέους και τις επιχειρήσεις. Έτσι μπορούν να ε, έχουν κάτι στα χέρια τους για να αξιολογήσουν, να αξιοποιήσουν τους νέους και πολλές φορές διστάζουν γιατί έχουν απλώς συγγραφικό στα χέρια μόνο. Οπότε να υπάρχει ένα σωστό feedback για το πώς ένας φοιτητής, ε, ένας, ένας νέος ε, συμπεριφέρεται στις πραγματικές συνθήκες και αυτό θα βοηθούσε πολύ. Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο, τα κρατημέλη και η Ευρώπη θα πρέπει να επενδύσουν στους νέους, να επενδύσουν σε τέτοια συστήματα. Συχνά σήμερα διαπιστώνουμε ότι μέσα στην κρίση οι πρώτες περικοπές που γίνονται στους προϋπολογισμούς είναι ε, ε, τα, κεφάλαια υπόρρη που αφορούν την εκπαίδευση των νέων. Οπότε να, αυτή σας η πρόταση είναι πολύ σωστή για αυτή τη διασύνδεση παιδείας απασχόλησης. Κύριε Αλτικλήβα, θέλουμε την αντίδρασή σα. Ευχαριστώ. Ε, είναι πολλέ ερωτήσει. Για να απαντήσω στην πρώτη σα ερώτηση. Εάν ε, μεσοπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα μάλλον μακροπρόθεσμα μπορούμε να προβλέψουμε ένα πρόγραμμα για τις ιδέες μας, να πω ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν επικεντρωθεί αρκετά στα μακροπρόθεσμο σκέλος του θέματος, τις μακροπρόθεσμες λύσεις. Τα μέτρα που έχουν λάβει ως τώρα είναι πολύ βραχίας ισχύως. Ένα παράδειγμα του είδους των μέτρων που μας λείπουν είναι ότι στη Σλοβενία λόγω χάρη δεν έχουμε στρατηγική για την ανεργία των νέων. Εάν υπήρχε μια τέτοια στρατηγική πριν από μια διετία, η τάση θα είχε ήδη μεταστραφεί. Είμαι υπέρ των μέτρων που είναι πιο διορατικά, με περισσότερο μακροπρόθεσμες επιδιώξεις, αλλά δεν ε, ε, υπάρχουν ακόμη. Στο δεύτερη ερώτησή σας να πω ότι βρίσκω περισσότερο σχολιασμό παρά ερώτηση. Τέλος πάντων συμφωνώ ότι ο τομέας της εκπαίδευσης και η έλλειψη συνδυασμού του εκπαιδευτικού χώρου με την αγορά εργασίας είναι ένα πρόβλημα. Είναι ελάχιστα τα παραδείγματα όπου οι εξετάσεις ε, και οι πρακτικές ασκήσεις δίνουν μόρια στους ε, νέους και αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Κοιτάξτε, εδώ έχετε ακούσει μάλλον ξανά για speed dating, ραντεβού express, αλλά όχι για ε, ακρόαση express. Τέλος πάντων καταφέραμε με, αυτό το, με αυτή τη μέθοδο να καλύψουμε πολλά διαφορετικά θέματα με μια ιδιαίτερη ματιά στις ανάγκες της ευρωπαϊκής νεολαίας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την ε, συμμετοχή σας και αυτό που ξέρω για το speed dating είναι ότι χτίζει κανείς, δημιουργεί καμιά φορά σχέσεις. Τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος το ραντεβού, έτσι, express. Ε, πάντως αυτό κάναμε και εμείς εδώ και αυτό κάναμε και το Μάιο όταν συναντηθήκαμε και θα ξαναβρεθούμε γιατί η σχέση μας θα κρατήσει στο χρόνο. Και εσείς και οι δικέ σα οι προτεραιότητε και οι μέρημνε θα είναι και δικέ μα. Σα ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Ε, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα άλλο συναρπαστικό θέμα, μια άλλη οδηγία. Ε, Τώρα έχουμε την πρόταση για πρόταση οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με του ναυτικού. Hm. Hm. Να προσθέσω ότι θέλω να ευχαριστήσω τους μεταφραστές, διότι αν υπάρχει ένα πρόβλημα στις ακροάσεις με συντομευμένες διαδικασίες είναι ότι δυσκολεύουμε πολύ τους δερμηνείς αλλά κάνατε πολύ καλή δουλειά οπότε θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς Uh, στην ημερήσια διάταξη τώρα, ανταλλαγή απόψεων για τους ναυτικούς. Ο λόγος στην κυρία Μωράν Σαρατιέ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που ευγενικά θα παραμένουν στην αίθουσα για αυτό το άκρο σημαντικό θέμα που θα έπρεπε να ενδιαφέρει όλα τα μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Γιατί είναι άκρο σημαντικό το ζήτημα αυτό. Διότι αγαπητοί συνάδελφοι, θα θυμάστε για όσους ήσασταν εδώ στην προηγούμενη θητεία, πρόκειται για μία και σχεδίου οδηγία, το οποίο είχε εγκαταληφθεί τον περασμένο Απρίλιο-Μάιο. Ε, ήταν πολύ περιορισμένος ο χρόνος που είχαμε. Γιατί μια νέα οδηγία για το θέμα αυτό. Διότι έχουμε όλοι μαζί υποχρέωση να ξαναδούμε κάποιες εξαιρέσεις που αφορούν τους ναυτιλωμένους και που θα έπρεπε να μας επιτρέψουν να ξαναδούμε τουλάχιστον πέντε οδηγίες. Αυτές που αφορούν την, ε, αυτή που αφορά την πτώχευση εταιριών, αυτή που αφορά την εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή που αφορά το δικαίωμα πληροφόρησης και διαβούλευσης ε, των ε, ναυτιλωμένων, την άλλη που αφορά τις συλλογικές απολύσεις, αλλά και τη μετατόπιση επιχειρήσεων καθώς και την απόσπαση εργαζομένων. Πρόκειται για θέματα Καθοριστική σημασία για την Επιτροπή απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων. Τη δουλειά αυτή πρέπει να την συνεχίσουμε λοιπόν, αλλά την συνεχίζουμε με μεγάλη διάθεση να πετύχουμε. Σε αυτό μας διευκολύνουν οι ακροάσεις που οργανώσαμε. Ακροάσεις για διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, με την Ομοσπονδία Ευρωπαίων Εργαζομένων και την Ευρωπαϊκή Ένωση Εφοπλιστών. Είμαστε, έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι η σύγκληση απόψεων σε κάποια θεμελιώδη σημεία θα μας εξυπηρετήσει στην συνέχεια της εξέτασης αυτής της οδηγίας. Το δεύτερο σημείο στο οποίο ήθελα να σταθώ είναι η μέθοδος εργασίας που θα ακολουθήσουμε. Πρέπει να ευχαριστήσω το σύνολο των σχεδόν εισηγητών, διότι ήδη μπορέσαμε να οργανώσουμε μία ε, συνεδρίαση για να τοποθετηθούν σε μια πρώτη φάση οι σχεδόν εισηγητές για τον τρόπο που θα εργαστούμε. Η δική μου πρόταση ήταν η εξής προσκάλεσα το σύνολο των πολιτικών ομάδων να έρθουν να συνεργαστούμε σε όλη τη διάρκεια επεξεργασίας του θέματος, ώστε να έχουμε τις ίδιες πληροφορίες συνέχεια, όλοι. Έτσι θα ε, είμαστε ε, σε ένα επίπεδο ε, ενημέρωσης κοινό. Ο καθένας μετά θα μπορεί να υποβάλει τις τροπολογίες που θέλει, αλλά θα έχουμε όλοι μαζί το ίδιο σύνολο πληροφοριών. Ως προς αυτό, νομίζω ότι και το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των πολιτικών ομάδων θα ωφεληθεί, αλλά και η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα της δουλειάς μας. Ο κοινό μας στόχος είναι προφανώς να πετύχουμε την αναθεώρηση του συνόλου αυτών των οδηγιών μέσω αυτής της αναθεώρησης οδηγίας για τους ναυτιλωμένους που θα λάβει σάρκα και οστά νόμοθετικός και όπως ήδη έχουν προλειάνει το έδαφος οι συνομιλίες μας με εφοπλιστές και ναυτιλωμένους, θα λάβουν λοιπόν σάρκα και οστά ε, με την σημαντικότατη ψηφοφορία που ελπίζουμε να συγκεντρώσει ευρύτατη πλειοψηφία στην Ολομέλεια. Και ενώ την προηγούμενη φορά η δουλειά μας έγινε υποπίεση χρονική λόγω των ευρωεκλογών που επίκυντο, τώρα βλέπουμε ότι έχουμε περισσότερο χρόνο. Βεβαίω και αυτό είναι σχετικό γιατί θα θέλαμε να καταλήξουμε σε ψηφοφορία στην Επιτροπή τον Μάρτιο και στην Ολομέλεια τον Απρίλιο ή Μάιο δεν έχουμε λοιπόν τόσο περισσότερο χρόνο, αλλά η δουλειά μας, εφόσον υπάρχει διαρκής αλληλενημέρωση των πολιτικών ομάδων, ίσως μας επιτρέψει να πετύχουμε. Σε κάθε περίπτωση, Πρόεδρε, να σας πω ότι ως εισηγήτρια είμαι απολύτως ε, αφοσιωμένη στην επίτευξη αίσιου πέρατος για την ε, έγκριση αυτής της ενωθέρωσης οδηγίας. Μαζί με τους συνεργάτες της γραμματείας που είναι καθισμένοι δίπλα σας και ελπίζω και με την συνεργασία όλων των σχεδόν εισηγητών για να έχουμε επιτυχία σε αυτό το κείμενο. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό όλοι μαζί να συνομιλούμε με τους ε, ενδιαφερομένους για το θέμα αυτό ε, όσους αφορά δηλαδή το θέμα, τους εφοπλιστές και τους ναυτιλωμένους. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Ο λόγος στην Κομισιόν. Κυρία Γκουίν. Πέντε λεπτά έχετε. Κυρία Γκουίν, το προφέρω σωστά το όνομά σας. Ναι, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η σημερινή συνεδρίαση αφορά την ακρόση σε συνάντηση με τους κοινωνικούς εταίρους. Οπότε και να δούμε τώρα ε, τι έγινε μετά τις εισηγήσεις ε, και θα σας μιλήσω μετά αφού ακούσουν τις γνώμες. Καλά λέει η Πρόεδρος. Μαρκ Ντίγκινσον τώρα. Από την Ομοσπονδία των εργαζομένων στις μεταφορές. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Συγγήτρια και αξιότιμοι βουλευτές. Όπως είπατε είμαι ο Μαρκ Ντίκινσον και είμαι ο Γενικός Γραμματέας αυτού του φορέα του Συνδικάτου των Εργαζομένων ε, στις θελάσσιες μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις κάτω Εδώ είμαι ε, ως εκπρόσωπος ε, αυτού του φορέα όπου και εξελέγει στα πλαίσια του γενικού διαλόγου για τις θελάσσιες μεταφορές. Επίσης είμαι αντιπρόεδρος της, της ETF για τις ε, μεταφορές. Όπως γνωρίζετε, η ETF είναι μία ένας φορέας. Ένας φορέας που αφορά τις μεταφορές και την αλία για τις μεταφορές. 213 213 είναι κατέχουμε σε 41 ευρωπαϊκές χώρες και βασούμε περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ερωσμένους στις μεταφορές, Όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές και υπερήφανα, εκφράζονται μέσω ημών 270.000 περίπου ε, σε 72 ε, συνδικάτα σε ένα σωρό χώρες, όπως είπαμε, για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου προσωπούμεθα και η αντιπροσωπευτικότητά μας όσον αφορά τα θαλάσσιες μεταφορές μαζί με τον ΕΞΑ είναι κάτι το αδιαμφισβήτητο. Και έτσι θεωρούμε λοιπόν ότι μπορούμε να έχουμε ένα συνεχιζόμενο διάλογο με τους εφοπλιστές εδώ και πολλές δεκαετίες. Και τώρα θα θέλαμε να σας δώσουμε το πλαίσιο αυτού του, αυτού του συμβασμού με την έξα, όσον αφορά τις εξαιρέσεις. Όπως γνωρίζετε, το κοινό ισχύει για όλους τους ε, κλάδους. Και μέχρι τώρα τα κράτη-μέλη μπορούσαν να προβλέψουν εξαιρέσεις για τους ναυτιλωμένους, για τους ναυτικούς, ε, λόγω της φύσης του τομέα των μεταφορών. Οπότε έτσι έχουμε διαφοροποιημένη μεταχείριση των ε, ναυτικών σε σχέση με τους εργαζομένους στις χερσές μεταφορές. Από πλευρά της Ομοσπονδίας μας, της ETF, αυτό είναι λάθος, πρέπει να διορθωθεί και με τρόπο αποτελεσματικό. Αυτό το οποίο τώρα αποσκοπούμε είναι το να τηρηθούν πάρα πολλά δικαιώματα τα οποία προβλέπονται από τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ισχύσουν αυτά τα δικαιώματα και για τους ε, ναυτικούς. Η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής που τροποποιεί τις σχετικές οδηγίες επομένως ήταν κάτι που το επιζητούσαμε και το περιμέναμε πώς και πώς. Βέβαια προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις υπέρ και κατά. Αλλά αν εξετάσει κανείς το πώς εφαρμόστηκε ήταν σαφές ότι προκλήθηκε κάποια σύγχυση και ότι δεν λύθηκαν πάρα πολύ βασικά μιλήματα των ε, κοινωνικών εταίρων. Να δούμε τώρα το ε, σημασία του γενικού διαλόγου. Οι γενικοί εταίροι τότε που εσείς ενταχθήκατε στο πρώτο μέτρο κατάλαβαν ότι θα πρέπει να γίνει ε, πιο, πιο νυφάλια συζήτηση και όχι τόσο φορτισμένη. Οπότε, η ETF και ο Φορέα των Φοντιστών είπαν να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσει τόσο ώστε να δούμε πού υπάρχει ένα κοινό παρονομαστή. Όπως λέμε και στην ε, Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου, ε, λέμε ότι μονός καυγάς δεν γίνεται και επομένως είπαμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε όπως και έγινε τόσα χρόνια βήμα-βήμα και γι' αυτό και σήμερα και εγώ, αλλά και η κυρία Βόση εδώ που κάθεται στα δράμα που έρχεται από την έξα, ε, μπορούμε να σας εκθέσουμε το συμβασμό, τη συμβαστική συμφωνία, να σας πούμε πού φτάσαμε συννοούμενοι όσον αφορά την υπόθεση αυτή της εξαίρεσης από κάποιων διατάξεων των ναυτικών. Οπότε, πρέπει να σας πω ότι ήταν ε, ευχάριστη έκπληξη το ότι συμφωνήσαμε. Δεν είναι κάτι που ήταν αυτονοητό την αρχή και αυτό που έκανε τη διαφορά ήταν το ότι η ETF και η ΕΞΑ είχαν δεσμευθεί να γίνει επικοδομητικός διάλογος και να γεφυρωθούν οι αρχικές διαφωνίες. Έτσι νομίζω θα γίνει πιο πρακτική η πρόταση της Επιτροπής. Όταν έρθει η ώρα να απολάβουν 100% τα δικαιώματά τους για πληροφόρηση και διαβούλευση ναυτική. Και επίσης όσον αφορά το δικαιωμά τους για δίκες και σωστές συνδικές εργασίες. Με την αδειά σας τώρα στην κυρία Βόσ θα δώσω το λόγο. Σου και αυτή δύο λόγια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Εισηγήτρια, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως είπε και ο Μάρκ, είμαι η Πία Βος, και είμαι πρόεδρος των εφοπλιστών στην Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εφοπλιστών ΕΞΑ για το γεγονός ότι μας προσκαλέσατε ως κοινωνικούς εταίρους για τις θαλάσσιες μεταφορές να παρουσιάσουμε την ε, κοινή μας συμφωνία επί των πέντε κοινωνικών οδηγιών. Η ΕΞΑ αντιπροσωπεύει τις Εθνικές Ενώσεις Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας. Οι εταιρείε μέλη των Εθνικών Ομοσπονδιών έχουν στο στόλο τους όλα τα είδη σκαφών και δραστηριοποιούνται σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι Ευρωπαίοι εφοπλιστές είναι πάρα πολύ δραστηροί τόσο στις παραδοσιακές εμπορικές μεταφορές αλλά και στην, στον υπεράκτιο, στις υπεράκτιες δραστηριότητε, όπου ε, διαθέτουμε υπερσύγχρονα σκάφη. Οι εφοπλιστές επίσης ασχολούνται τόσο με τις επιβατικές μεταφορές και τις μεταφορές αγωθών. Είτε μιλάμε για κοντέινερ είτε για box. Τέλος, οι εφοπλιστές δεν δραστηριοποιούνται μόνο σε εμπορικές συναλλαγές από και προς ευρωπαϊκά λιμάνια. Το ίδιο κάνουν και σε ε, εμπορικές συναλλαγές μικρών αποστάσεων, σε γειτονικές χώρες, σε Ευρωπαϊ... στην... Ε, γειτονικές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε διατλαντικές μεταφορές. Επίσης, οι εφοπλιστές συμμετέχουν και σε εμπορικές συναλλαγές εκτός Ευρωπαϊκής Υπήρου. Μια πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου της Οξφόρδης υπέδειξε ότι οι Ευρωπαίοι εφοπλιστές ελέγχουν το 40% του παγκόσμιου στόλου βάσει χωρητικότητας και έχουν εργαζόμενους 2,3 εκατομμύρια ανθρώπους. Η συνεισφορά στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ είναι περίπου 145 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή η οικονομική πραγματικότητα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν συζητούμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, πρόταση οδηγίας για την κατάργηση των εξαιρέσεων που ισχύουν για τους ναυτικούς. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε το γεγονός ότι το θέμα αυτό δεν είναι απλά ένα απλό, μια απλή διοικητικού χαρακτήρα τροποποίηση πέντε σχετικών οδηγιών. Κάθε άλλο. Πρόκειται για ένα περίπλοκο ζήτημα, τόσο από νομική σκοπιάς, όσο και αν λάβει κανείς υπόψη τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για τον ευρωπαϊκό εφοπλισμό και τους ευρωπαίους ναυτικούς. Με άλλα λόγια, οι συζητήσεις μεταξύ της ΕΞΑ και του ETF για το ζήτημα αυτό ήταν κάθε άλλο παρά μια εύκολη διαδικασία. Το αντίθετο, χρειάστηκε πολύς χρόνος για να κατανοηθεί η περιπλοκότητα του ζητήματος και να εξοικειωθούμε ε, η κάθε πλευρά με τα συμφέροντα και τους προβληματισμούς της άλλης. Παρ' όλα αυτά, παρά τις πολύ δύσκολες συζητήσεις που είχαμε, η ΕΞΑ και το ETF κατάφεραν να κάνουν αυτό που πολλοί θα θεωρούσαν αδύνατο. Καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με συγκεκριμένες προτάσεις για την τροποποίηση της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κοινή μας πρόταση αντιπροσωπεύει αυτό που λέω που ονομάζω εγώ δίκαιη αλλά και λεπτή ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των δύο οργανώσεων και η πρόταση αυτή τη χάνει της έγκρισης των μελών των οργανώσεών μας. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, το, η περιπλοκότητα του ζητήματος έχει πλέον αναγνωριστεί από όλους τους εμπλεκόμενους από την ΕΞΑ και το ETF και τα μέλη τους, αλλά πιστεύω επίσης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιο πρόσφατα από το Συμβούλιο των Υπουργών. Ελπίζουμε ότι και εσείς θα αναγνωρίσετε την περιπλοκότητα στις επικείμενες συζητήσεις που θα έχετε για το θέμα και ότι θα λάβετε υπόψη σας το γεγονός ότι οι κοινωνικοί εταίροι έχουν καταλήξει σε μια δίκαιη αλλά λεπτή και ισορροπημένη συμφωνία. Μια συμβαστική πρόταση ή όπως είπε και ο Μάρκ καταφέραμε να χορέψουμε ταγκό. Ευχαριστούμε. Και τώρα να δώσω το λόγο στους σκιώδεις ασυγητές. Μερικοί είναι εδώ στο Προεδρείο. Να δώσω το λόγο στην Άγνες Γιονκέριους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτούς που σήμερα ε, είναι εδώ. Ιδίως τους εκπροσώπους της Επιτροπής που μας εξηγούν τη σημασία επίτευξης συμφωνίας και γι' αυτό να σας ευχαριστήσω πρώτα-πρώτα. Δεν ήταν τίποτα το διασκεδαστικό, δεν ήταν ένας περίπατος στο πάρκο, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, αλλά... Εδώ πέρα Καταλαβαίνουμε ότι ε, κάνατε μεγάλες προσπάθειες και γι' αυτό πρέπει να σας συγχαρούμε. Αλλά για τους κοινωνικούς τέρους και μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια διαδρομή που την έχουμε γνωρίσει και από άλλες περιπτώσεις και επειδή η συμφωνία αυτή και οι τομεακές ε, συμφωνίες είναι πολύ σημαντικές. Εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα, εκείνοι που τις έχουν συνάψει γνωρίζουν καλύτερα τα δικαιώματα και τις ανάγκες των αυτιλωμένων. Σε ευρωπαϊκό λοιπόν επίπεδο Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να επιληφθεί το Ευρωκοινοβούλιο γιατί αυτή είναι η καλύτερη λύση και έπειτα για το ίδιο το περιεχόμενο του κειμένου πρέπει να είναι πολύ σαφές. Και καταλαβαίνω ότι έχουν γίνει πολλές συζητήσει ε, την τελευταία στιγμή για πολλά διαφορετικά σημεία. Μπορείτε να μας πείτε ποια ήταν αυτά τα αμφιλεγόμενα σημεία. Και κάτι άλλο που το ρωτάω από καθαρή περιέργεια. Γιατί για τους ναυτιλωμένους προβλέψατε να μιλήσετε μόνον για τους ε, αρμόδιους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί περιοριστήκατε μόνο στους ευρωπαϊκούς φορείς. Και η ερώτησή μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η εξής. Νομίζω το είπε η κυρία Βός μιλήσαμε για τη θετική αποδοχή της πρότασης αυτής από το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Η Επιτροπή μπορεί να μας το επιβεβαιώσει ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή ταυτίζονται στις απόψεις τους για τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσαμε να προωθήσουμε το θέμα αυτό. Δηλαδή η τομεακή συμφωνία να ε, χρησιμοποιηθεί ως βάση. Ευχαριστούμε η κυρία Τούρνες. Øh, Ευχαριστώ. Και εγώ να ευχαριστήσω όλου του προσώπου των κοινωνικών εταιρεών και κατέφεραν πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια. Προέρχομαι από την Δανία και ακριβώ γι' αυτό το λόγο είμαι εξοικειωμένη στο ότι όταν οι συνομιλούντες τα βρίσκουν είναι υποχρεωμένοι οι πολιτικοί να σεβαστούν την συναυθήσα συμφωνία. Οπότε αυτό που θέλω να ρωτήσω αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα με ενδιέφερε να μας πείτε πώς αξιολογείται αυτή τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων. Είναι αυτό το οποίο εσείς επιζητούσατε από την αρχή. Μας είπαν ότι χρειαζόταν να υπάρξουν υποχωρήσεις άλλος εδώ, άλλος εκεί, ούτως ώστε να καταλήξουν συμφωνία. Φαντάζομαι δε ότι και εσείς θα πρέπει βέβαια να κάνετε κάποιες μικροπόσαρμογέ και γι' αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον να μας πείτε τη γνώμη σας. Σε σχέση με αυτό που ακούσαμε τους χιονικού εταίρους. Thank you. Uh, not here. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι εδώ η Άννα Γκερίκη. κυρία Μάκιντάιρ. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι αλήθεια, η Άννα και δεν μπορούσε να είναι εδώ, οπότε μου ζήτησε να πω κάποια λόγια εκ μέρου του ECR. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους ομιλητές. Να ευχαριστήσω και την εισηγήτριά μας, διότι η κυρία Σαρτία πάντοτε κάνει καλή δουλειά για την Επιτροπή μας και νομίζω ότι δεν θα αποτελέσει εξαίρεση η συγκεκριμένη δουλειά της. Η παγκόσμια φύση των θαλάσσιων μεταφορών και η προσπάθεια να αναζητηθεί ποιο έχει τη δικαιοδοσία καθιστά την εφαρμογή της νομοθεσίας σε εθνικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο πολύ δύσκολη υπόθεση. Το ECR χαιρετίζει λοιπόν την πρόταση της ε, Κομισιόν για την τροποποίηση της οδηγίας. Φάνηκε ότι θα, υπήρχε πολύ, θα υπήρχαν πολύ μικρά ωφέλη από την οδηγία. Θα χρειάζονταν μεγάλες τροποποίησεις και μια, ε, ένας εκ νέου ορισμός των βασικών θεμάτων. Επίσης δεχόμαστε ότι το τρέχον σενάριο είναι θετικό. Γι' αυτό μπορούμε να ε, αποδεχθούμε την εξαίρεση των ε, ναυτικών. Η βασική ανησυχία είναι ότι οι εφορπλιστικές εταιρείε προσπαθούν να αποκτήσουν νέες ε, σημαίες και έτσι ενδεχομένως να έχουμε απώλειες. Οι ενδείξεις μας από τους κοινωνικούς εταίρους δείχνουν επίσης ότι αν η οδηγία αναγνωρίσει τις μοναδικές συνθήκες εργασίας των ε, ναυτικών θα μπορούσαν οι αλλαγές να γίνουν με πολύ μικρό κόστος όσον αφορά τις ε, δραστηριότητες. Τα συνδικάτα καλούσαν πάντοτε την, ε, να διευκολύνουν ε, την ε, επιβολή της πρότασης. Στην μελέτη επιπτώσεων της Κομισιόν δεν φαίνεται να υπάρχουν ενδεχόμενα κόστη. Στατιστικά δεδομένα δεν υπάρχουν για τους ναυτικούς. Παρ' όλα αυτά η Κομισιόν εκτιμά ότι όσον αφορά η την ε, επικοινωνία EWC θα μπορούσε το κόστος να ανέλθει σε 635 ευρώ αναμέλως ανασυνάντηση. Συμπερασματικά λοιπόν υπάρχει γενική συμφωνία ότι μόνο η ευρωπαϊκή νομοθεσία μπορεί να δημιουργήσει ένα μορμονισμένο καθεστώς για τα δικαιώματα των ναυτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, ως πολιτική ομάδα έχουμε τους προβληματισμούς μας και νομίζουμε ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν νέα βάρη που πολύ λίγα ωφέλη θα επιφέρουν στην όλη κατάσταση. Ευχαριστώ. Ο Πάτρικ Λιάρη δεν είναι εδώ. Τζιν Λάμπερτ δεν είναι εδώ επίσης. Τότε ο λόγος στην κυρία Αγιούτου Ντανιέλα εκ μέρους του, της ομάδας EFDD. Ευχαριστώ πρόεδρε συνάδελφοι. Σήμερα αντικαθιστώ τη συνάδελφο Τιτσιάνα Μπεγκίν που είναι η σκιώδης εισηγήτρια για αυτή την πρόταση. Δεν μπορούσε όμως να είναι εδώ γιατί έχει ανελημμένες υποχρέωσεις στη Ρώμη. Βλέπουμε πολύ θετικά την πρόταση της Επιτροπής διότι έχουν δικαίωμα μεγαλύτερης κοινωνικής προστασίας συναυτιλόμενοι από ότι άλλες κοινωνικές κατηγορίες. Θα πρέπει λοιπόν να προβλεφθεί κάτι τέτοιο, διότι η χαμηλή κοινωνική προστασία έχει κάνει λιγότερο ελκυστικέ τι θέσει εργασία στα επαγγέλματα τη ναυτιλία. Ιδίω ε, η έλλειψη εργατικού δυναμικού και χαμηλότερων προσόντων είναι κάτι που ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αισθητό. Γι' αυτό καλωσορίζουμε και τη συμμετοχή στην επίτευξη συμφωνία όλων των κοινωνικών συνομιλητών και είναι ένα τομέα που χρειάζεται σαφώ την δική μα στήριξη. Υποδεχόμαστε θετικά την πρόταση οδηγία, ευχαριστούμε την εισηγήτρια και θα θέλαμε να συνεργαστούμε με τους υπόλοιπους συναδέλφους για να είναι γρήγορη η εξέταση του θέματος με αίσιο αποτέλεσμα, ακολουθώντας και τις προτροπές και τις συμβουλές των κοινωνικών εταίρων. Uh, uh, Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στην κυρία Νίριαντ, Άντ, η οποία εκπροσωπεί την Επιτροπή Αλίας Ευχαριστώ. Νομίζω ότι βρισκόμαστε όλοι στην ίδια θέση εδώ ως προς την... Ε, και έχουμε την ίδια άποψη για, την... για το ιδιαίτερο βάρος και τις ίδρες ανάγκες των αυτιλωμένων. Γι' αυτό καλωσορίζουμε την πρόταση της Επιτροπής. Πρέπει να προβλέψουμε περισσότερη ασφάλεια και προστασία για αυτούς τους ανθρώπους εργαζομένους και να ε, έχουμε ένα αίσιο πέρα στο γραφειοκρατικό άχθος που αυτή τη στιγμή τους επιβαρύνει, αλλά να αντιμετωπίσουμε και το κοινωνικό dumping η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλώ αναγνωρίζει το κοινωνικό ντάμπινγκ σε αυτόν τον τομέα και γι' αυτό σωστά συμπεριλαμβάνει την ρήτρα μη ε, υπαναχώρηση και τη σταδιακή μείωση. Όμω για τι ε, συλλογικέ απολύσει, οι κοινοποίηση πιστεύουν δεν θα πρέπει να γίνονται στι αρμοδείς αρχέ του κράτου σημαία μόνον, αλλά να συμπεριλαμβάνεται και το κράτο όπου προσλήφθηκαν οι εργαζόμενοι εφόσον είναι διαφορετικό. Επίση, η δυνατότητα εξαίρεση από τι υποχρεώσει συλλογικών απολύσεων εφόσον μιλάμε για ένα και μόνο σκάφο, Αυτό θα πρέπει να αφορά συγκεκριμένα σκάφη, γιατί ξέρουμε ότι το μέγεθο και οι διαστάσει του, καθώ και ο αριθμό του πληρώματο που απασχολούν, ε, είναι πολύ διαφορετικό. Δεν μπορούμε να έχουμε μία κοινή λύση για όλους. Ε, θα πρέπει να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση ανάλογα με το αν μιλάμε για ένα μεγάλο σκάφος ή κάποιο με οικογενειακό πλήρωμα που είναι μια, μέλη μια οικογένεια. Επίση, για του αλληλεί θα πρέπει να προσφέρουμε ένα σοβαρό επίπεδο προστασία σε όλη τη διάρκεια τη ταδιοδρομία του, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια και στην απασχόλησή του για όλου του εργαζομένου το τομέα. Διότι ξέρουν ότι, θα πρέπει να ξέρουν ότι όσο ε, μεγαλώνουν θα μπορούν να έχουν ενεργό ρόλο στην αγορά εργασία αυτή. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να είναι ε, συνεπέ και να συνάδει με τι προτεραιότητέ μα για την απασχόληση και τι νέε θέσει εργασία. Θα πρέπει οι κοινότητε των αλλιών να προστατευτούν και να βελτιωθεί το κύρο του τομέα τη ναυτιλία. Υπάρχουν βεβαίω κάποιε ανησυχίε για τον τεχνικό εξυγχρονισμό και το κόστο που μπορεί να επιφέρει. Γι' αυτό ως μέλος της Επιτροπής Αλίας πιστεύω ότι μπορούμε να προβλέψουμε μια σχετική σύσταση που ενδεχομένως να προβλέψουν περαιτέρω κονδύλια. Κονδύλια για τα σκάφη που χρειάζονται βελτίωση εξυγχρονισμού του εξοπλισμού τους για να συνεχίσουν να λειτουργούν σωστά. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιοποιήσει το δυναμικό που υπάρχει εδώ, καθώ και όλε τι δυνατότητε των νεαρών αλλιέων. Έχω και μια ερώτηση. Αναφέρατε την ε, μελέτη δικτύπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα εξαχθούν δύο μελέτε. Μία για την αλλαγή σημαία και μία για την ε, ε, φάση ύφεση και, και υποβάθμιση τέλους μάλλον, της αδειοδομία των αλλιέων. Ε, ήθελα να μου πείτε τι πιστεύετε ότι θα λάβετε ως πόρισμα από τις δύο αυτές μελέτες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Και τώρα λόγω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποιε ερωτήσει και παρατηρήσει για το θέμα αυτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτές οι συζητούμενες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζητώνται σήμερα και δεν έρχονται από το πουθενά. Εδώ και πολλά χρόνια τις εκπονούμε. Να σας υπενθυμίσω το ιστορικό πλαίσιο, όπως κάθε πρόταση στο πλαίσιο του άρθρου 153 της συνθήκης όσον αφορά το κεφάλαιο για την κοινωνική πολιτική εμείς καταθέτουμε τις προτάσεις μας μόνο αφού έχουμε διεξαγάγει κάποιες ε, διαβουλεύσεις του άρθρου 154 με τους κοινωνικούς εταίρους. Παίρνουμε δύο φάσεις διαβούλευσης. Και τότε κοινωνικοί εταίροι για την Αλία είχαν εγκρίνει την πρότασή μας να μπει τέλος στις εξαιρέσεις ε, όσον αφορά αυτές τις ε, οδηγίες και όσον αφορά τους ναυτιλωμένους τότε οι χιονικοί δεν είχαν συμφωνήσει. Ήταν θετικά τα συνδικάτα αλλά οι εργοδότες όχι. Και δεν έγιναν τα πράγματα ακριβώ όπως τα είχαμε ζητήσει τότε ως διαπραγματεύσει και γι' αυτό και εμείς συγχαρητήσαμε την αξιολόγηση των επιπτώσεων και Συνεχίσαμε επίσης και τον διάλογο με τους χιονικούς εταίρους. Για να μπορέσουμε να εξετάσουμε αυτές τις ιδιοτυπίες που αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν στον κλάδο. Οπότε και στις ε, προτάσεις μας προσπαθήσουμε να έχουμε ένα πλαίσιο ώστε να απαλλάξουμε από το οικονομικό βάρος των αλλαγών. Επίσης είχαμε μία προσέγγιση φιλόδοξη, ούτω ώστε να έχουμε σύγκληση και προσέγγιση των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των εργαζομένων στη θάλασσα. Και από τον Νοέμβριο του 2013 οι επαφές με τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο κατέδειξαν ότι κάποια κράτη-μέλη που έχουν κλάδο ε, ιδιαίτερα εκτεταμένο όσον αφορά ε, της, τη ε, θαλάσσια οικονομία και συναντήθηκαν οι κοινωνικοί εταίροι όταν διαπιστώθηκε ότι κάποιες προτάσεις της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν συγκέντρωναν μετά από συζητήσεις τη Συμφωνία των Μέλων του Συμβουλίου. Ναι, είπαμε ότι χρειάζονται δύο τα γκόρ και μονός καυγάς δεν γίνεται, αλλά ε, είπαμε ότι για τις συνομοθέτες πρέπει να συμφωνήσουν. Αλλά και εμείς με τη σειρά μας θεωρήσαμε ότι είναι πάρα πολύ θετικό τότε συμφώνησαν με τις συνομιλίες τους οι κοινωνικοί εταίροι και έτσι φτάσανε σε κάποια λύση. Οπότε και συνεχίστηκαν οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο. Η αξιολόγηση που κάνουμε τώρα είναι το ότι οι κοινωνικοί εταίροι συμφωνούν με τους γενικούς στόχους της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως, παρ' όλα αυτά, οι κοινωνικοί εταίροι βρήκαν μια διαφορετική ισορροπία σε κάποιες διατάξεις από τα όσα είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως, πρέπει να δούμε τώρα το σύνολο και την συνολική ισορροπία και να υπογραμμίσουμε το ότι έχουμε τους ίδιους γενικούς στόχους. Προχωρούν περισσότερο σε κάποια σημεία κοινωνική εταίροι, ε, σε άλλα προχωρά περισσότερο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε κανείς θα πρέπει να εξετάζει το σύνολο. Και όσον αφορά τις συζητήσεις στο Συμβούλιο, η συνεννόηση των κοινωνικών εταίρων θεωρήθηκε κάτι το χρήσιμο, κάτι το θετικό από μία σειρά κρατημέλια. Από πλευρά μας δε μείναμε σταθεροί σε απόψεις μας γιατί μιλούμε για ε, συνομοθεσία και τις επόμενες εβδομάδες Συμβούλιο και Κοινοβούλιο πρέπει να συμφωνήσουν αρχές του 2015. Τώρα για να απαντήσουμε σε κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις απλώς να σας πω το εξής. Κύριε Μακιντάρη νομίζω ρώτησε για την αξιολόγηση ε, των επιπτώσεων και όσον αφορά το κόστος των αλλαγών που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλάμε για τη σελίδα 39 αυτής αξιολόγησης. Εκεί έχουμε και την αξιολόγηση του κόστους για τις αλλαγές όσον αφορά την κατάρτιση και την ενημέρωση. Εδώ θα πρέπει να κοιτάξουμε κάποιες δαπάνες όλα αυτά στην εξηγήση των επιπτώσεων τη δική μας. Κυρία Συγκίτρια, έχει κάποιε άλλες συγκεκριμένε παρατηρήσει. αλλά θα τι απαντήσω στην Επιτροπή Ελίας μεθαύριο. Uh, Ευχαριστώ, Μάρκ Ντίκινσον. Έχετε λίγα λεπτά για να συνοψίσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να επανέλθω στο προφανές ερώτημα που έθεσε ο σκιώδης εισηγητής, η σκιώδης που ρώτησε αν οι κοινωνικοί εταίροι θέλουν την υποστήριξή σας. Βεβαίως και τη θέλουμε και τη χρειαζόμαστε. Η συμβιβαστική μας πρόταση φυσικά δεν είναι δεσμευτική αλλά θα τολμήσω να προτείνω ότι με αυτόν τον τρόπο πρέπει να ειδωθεί η συμφωνία. Πρέπει να θεωρηθεί ως ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα και καταδεικνύει την ανάγκη να υπάρχει ένας ενεργός και επικοδομητικός κοινωνικός διάλογος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και γνωρίζουμε ότι η Κομισιόν εναποθέτει μεγάλες ελπίδες στην πρακτική του κοινωνικού διαλόγου και η δική μου οργάνωση, αλλά θεωρώ ότι και οι συνάδελφοι μου από την έξα συμφωνούμε. Η συμβαστική μας πρόταση δεν είναι τέλεια, αλλά κανένα συμβασμός δεν είναι ποτέ τέλειος. Καταφέραμε να συμφωνήσουμε όσον αφορά την ε, κατάργηση των εξαιρέσεων και την ίση μεταχείριση των ναυτικών με τους ε, εργαζόμενους στη στεριά και καταφέραμε να βρούμε λύσεις σε πολύ ευαίσθητα ζητήματα όπως εξήγησε και η Πία στην παρέμβασή της, καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια πολύ λεπτή ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των δύο οργανώσεων, αλλά είναι ο καλύτερος συμβιβασμός στον οποίο μπορούσαμε να καταλήξουμε. Και από αυτή την άποψη θα θέλαμε να καλέσουμε όλους να λάβουν υπόψη τους πολύ σοβαρά στις συζητήσεις που θα γίνουν την πρότασή μας γιατί θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα ε, θετικό αποτέλεσμα τόσο για τους Ευρωπαίους ναυτικούς όσο και για τους Ευρωπαίους εφοπλιστές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Βός. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τον Μαρκ Δίκινσον όσον αφορά τη φύση της συμφωνίας μας. Και παρότι δεν θεωρείται δεσμευτικού χαρακτήρα συμφωνία μεταξύ κοινών εταιρεών. Εμείς τη θεωρούμε ως τέτοια, ως δεσμευτική συμφωνία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να απαντήσω σε ένα ερώτημα της σκιώδους Συγκίδριας που σχετιζόταν με τις συλλογικές απολύσεις. Η αξίζει να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν, η ΕΞΑ και το ETF έχουν συμφωνήσει να εφαρμόσουν την οδηγία για τις συλλογικές απολύσεις στην, ε, ε, στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών. Σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή συλλογική ε, απόλυση, ακολουθούνται οι διατάξεις της σχετικής οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής περίοδου που προβλέπεται. Θα πρέπει δηλαδή όλα τα μέρη να περιμένουν 30 μέρες έως ότου εκτελεστεί το σχέδιο απολύσεων. Και σε αυτή την περίοδο μπορούν τα πράγματα να ηρεμήσουν και να εξευρεθούν λύσεις μεταξύ του εργοδότη και των ε, εργαζομένων όσον αφορά τις συλλογικέ ε, απολύσεις. Και όταν διεξάγονται συλλογικές απολύσεις, οι αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας θα πρέπει να, να ενημερώνονται για την απόφαση αυτή. Και αυτό προβλέπεται στην οδηγία. Και η αρχή της, ε, του κράτους σημαίας ακολουθείται σε πάρα πολλά κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε. Κυρία Μωρέν Σαρτιέ, έχετε το λόγο για μια τελευταία παρέμβαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τους ε, συνομιλητές μας οι οποίοι συμμετείχαν στην ε, παρουσίαση της σημασία του θέματος αυτού για την Ευρώπη. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για την ευρωπαϊκή οικονομία και είναι πολύ σημαντικές οι οδηγίες που επιτέλους πρέπει να εξυγχρονιστούν. Και αυτό για να φύγουμε από το πρόβλημα των εξαιρέσεων και των αποκλεισμών. Δεύτερον, και αυτό ε, με ενδιαφέρει ιδιαίτερος προσωπικά, είναι η σημασία αυτής της προκαταρκτικής συμφωνίας που έγινε μέσω των διαβουλεύσεων δεν υποτιμώ καθόλου το σημαντικό αυτό αποτέλεσμα, όμως σίγουρα πρέπει να υπάρξει και μια κοινή συνειδητοποίηση της σημασία του θέματος μετά την αποτυχία υλοποίησης του της πρώτης απόπειρας ε, αναθεώρησης της οδηγίας τον περασμένο Μάρτιο-Απρίλιο. Νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό η αποτυχία αυτή, η έλλειψη αποτελέσματος, τελικά έφερε και κάτι θετικό. Μας κινητοποίησε όλους και από τη δική σας πλευρά και από τη δική μας, από την πλευρά του Κοινοβουλίου για να πετύχουμε επιτέλους αυτή τη φορά. Δεν έχουμε επιτέλους το δικαίωμα να αποτύχουμε. Γι' αυτό σε συνεργασία με τους σχεώδεις φυσικητές όλων των πολιτικών ομάδων Πρώτα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια κοινή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και μετά σε όλες τις υπόλοιπες κινήσεις μας. Το τρίτο σημείο στο οποίο θα ήθελα να εμείνω και επειδή το είπατε και πολλοί από εσάς είναι η σημασία των όσων προκύπτουν από τον κοινωνικό διάλογο. Σας, ε, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ως προς αυτό και μάλιστα συμφωνώ τόσο που πρότεινα στο σύνολο των συναδέλφων, των σχεδόν εισηγητών ε, των διαφορών πολιτικών ομάδων μέσα σε μία ομάδα διακομματική όπου έχουμε εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων και βουλευτές τα με, μεταξύ των μελών. Σε αυτή λοιπόν διακομματική ομάδα θέλουμε να περάσει το θέμα αυτό, διότι θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι θα πετύχουμε την ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία και τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση στην Ολομέλεια. Πρόκειται για ένα θέμα που μου φαίνεται ιδιαίτερος σημαντικό. Νομίζω το είπατε. Είναι περίπλοκο το θέμα. Έχετε κάνει πολλή δουλειά. Τη σέβομαι. Αλλά απευθύνω έκκληση στο σύνολο των συναδέλφων και σχεδόν εισηγητών στο βαθμό όπου υπάρχουν ε, διαφορετικές οδηγίες που αφορά το θέμα αυτό, πέντε έτσι, το είπα και προηγουμένως, θα πρέπει το Κοινοβούλιο να κάνει πραγματικά τη δουλειά του ως νομοθέτης εδώ. Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι το να διορθώνει κανείς οδηγίες σημαίνει ότι αναλαμβάνουν ε, οι γλωσσομαθείς νομική, υπάρχει μεγάλο επίπεδο λεπτομέρειας και εξειδίκευσης, είναι πολύ σημαντικό να κάνει κανείς ακριβώς αυτό, να νομοθετήσει. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το δει κανεί ε, συνολικά, σαν δέσμη πακέτο, αλλά βάσει τη συμφωνίας που έχετε για την εργασία των αυτιλωμένων και με όλους τους ενδιαφερόμενους και εμείς στο επίπεδο του Ευρωκοινοβουλίου πρέπει να κάνουμε τη δική μας νομοθετική ε, δουλειά και φαντάζομαι ότι θα μπορούμε να υπολογίζουμε στη συνεργασία των ΜΕΝ και των ΔΕ. Πάντως με αυτή την νομοθετική διαδικασία ελπίζω ε, να συμφωνήσουμε και μιλάω στο πρώτο πληθυντικό διότι όλοι συμμετέχουμε εδώ και να λάβουμε αποφάσεις που να συνάδουν με τη Χάρτα Θεμελιδών Δικαιωμάτων που εγκρίναμε. Δεν υπάρχει λόγος ως νομοθέτες από τη μια να εγκρίνουμε μια Χάρτα Θεμελιδών Δικαιωμάτων και μετά να αρκούμαστε σε αποκλεισμούς ή εξαιρέσεις της μιας της άλλης κατηγορίας εργαζομένων. Και ακόμη δύο λόγια, αν μου επιτρέπετε, θέλουμε πραγματικά οι νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ήδη σε κάποια σκάφη, ε, έφυγε συνάδελφος της Επιτροπής Αλίας, αλλά από αύριο μπορεί να χρησιμοποιούνται και από αλλιευτικά σκάφη. Έφυγε, αλλά ελπίζω θα τις μεταφερθούν αυτά που λέμε εδώ. Οπότε εδώ καλό είναι να γνωρίζει και το πλήρωμα το τι θα συμβεί. Σήμερα υπάρχουν πολλοί τρόποι να ε, έχουμε και την άποψη του ε, επαγγελματικού κλάδου. πολύ γρήγορα ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα όπως το αντιλαμβανόμαστε τώρα βάσει του προγραμματός μας. Σήμερα με την συζήτηση αυτή ξεκινούμε τις εργασίες μας εδώ στην Επιτροπή αλλά ήδη έχουμε συναντηθεί σε επίπεδο πολιτικών ομάδων. Έχουμε προετοιμάσει ένα πρώτο σχέδιο κειμένου που θα αποσταλεί στις μεταφραστικές υπηρεσίες με ε, προθεσμία της 18 Δεκεμβρίου. Βλέπετε πόσο γρήγορα πάνε τα πράγματα. Και θα εξετάσουμε αυτό το σχέδιο έκθεσης στην συνεδρίασή μας, κυρία Πρόεδρε, στις 21 ή 22 Ιανουαρίου 2015. Ελπίζουμε έτσι να φτάσουμε σε, στις 29 Ιανουαρίου με τη λήξη υποβολής, της διορίας για την υποβολή τροπολογιών θα εξετάσουμε τις τροπολογίες αυτές στις 26 Φεβρουαρίου και θα κοιτάξουμε μεταξύ των σκιωδών εισηγητών να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες τις εβδομάδες 10, 11 ή 12 ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ψηφοφορία χωρίς δυσκολίες στην Επιτροπή Απασχόλησης και ξέρετε ότι δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τη σημασία της ψηφοφορίας στην Επιτροπή. Ε. Ξέρετε ότι η σημασία αυτή και ο βαθμός στήριξης της πρότασης στην Επιτροπή Απασχόλησης θα εξαρτηθεί και θα καθορίσει την επιτυχία της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια. Ελπίζω λοιπόν ότι μπορώ να υπολογίζω σε εσά και μπορείτε κι εσείς να υπολογίζετε στην πλήρη αφοσίωσή μου για την επιτυχία αυτής της οδηγίας. Ευχαριστώ όλους και ελπίζω να έχουμε ένα αγαστό πνεύμα συνεργασίας για όσους κάθονται γύρω μου. Thank you and the... Ευχαριστώ έγκριση στην Επιτροπή Απασχόλησης έχει προγραμματιστεί για 24 Μαρτίου. Ευχαριστώ όλους όσους παρενέβησαν. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τριών λεπτών προτού προχωρήσουμε στη συζήτηση για το Γιούρες. Uh, uh, Ωραία, ξεκινάμε με το θέμα της μίλησης διάταξης για το EURES, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υπηρεσιών Απασχόλησης, πρόσβαση των εργαζομένων στις υπηρεσίες της κινητικότητας και περαιτέρω ολοκλήρωση των αγορών εργασίας. Κάθε ομιλητής που θα λάβει το λόγο θα έχει έξι λεπτά για την παρουσίασή του. Πρώτος είναι ο κύριος Ρόμπερτ Πλούμερ από την Eurobusiness. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να σας υποβάλω κάποια σχόλια εκ μέρους της Business Europe. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να πω ότι υποστηρίζουμε τα μέτρα που μπορούν να, προσ... προωθήσουν την κινητικότητα μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών και θεωρούμε ότι το Euros μπορεί να διαδραματίσει έναν ιδιαίτερα, ιδιαίτερο ρόλο ιδιαίτερα όσον αφορά το στόχο της οδηγίας για, την, για τον εξοχρονισμό του γιούρες και την καλύτερη αντιστοίχηση της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα πρέπει να υπογρομίσουμε ότι είναι σημαντικό ότι οι εργοδότες διατηρούν σημαντική ευελιξία όσον αφορά τη δυνατότητά τους να εξαιρούν θέσεις απασχόλησης που προκυρήσουν ε, από το Γιώρες και αυτό αφορά και την, τον, το νέο πεδίο εφαρμογή του Γιώρες που θα αφορά και τη συμπερίληψη των ιδιωτικών εργοδοτών και τις διασυνοριακές πρακτικές ασκήσεις. Υποστηρίζουμε αυτές τις ε, διαστάσεις επί της αρχής, αλλά υπάρχουν και κάποια πιο συγκεκριμένα θέματα στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ επίσης. Όπως είπα, υποστηρίζουμε την αρχή που σχετίζεται με τις πρακτικές ασκήσεις. Θεωρούμε ότι μπορούν αυτά να ενισχύσουν την απασχολησιμότητα των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα και μπορούν να προσφέρουν και ορισμένα πλεονεκτήματα στους εργοδότες. Σε σχέση με αυτό και ιδιαίτερα όσον αφορά τις πρακτικές ασκήσεις, Υπάρχει ένα θέμα στο οποίο θέλω να αναφερθώ, το οποίο είναι ζήτημα αρχής και αφορά τον ορισμό των πρακτικών ασκήσεων στον ε, κανονισμό, όπου αναφέρεται ότι οι πρακτικές ασκήσεις θα, οδηγήσουν, ε, θα θεωρηθούν ε, απασχόληση και εμείς Θέλουμε να πούμε ότι δεν θεωρούμε ότι οι πρακτικές ασκήσεις οι ασκούμενοι είναι εργαζόμενοι και αυτό είναι ένα σχόλιο για το άρθρο 2, το άρθρο με τους ορισμούς. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει περιθώριο στον κανονισμό να αναγνωρίζονται τα διαφορετικά καθεστώτα των ασκουμένων. Επίσης, ο κανονισμός ευθύνεται, ε, απευθύνεται κυρίως ε, στην αγορά εκπαιδευτικών ε, πρακτικών ασκήσεων όσον αφορά τα, τα διασυνοριακά υπάρχει και εξαίρεση των ε, πρακτικών ασκήσεων αλλά αυτό που θέλουμε να θέσουμε εμεί είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των προγραμμάτων Erasmus και Eures. Βλέπουμε ότι το Erasmus προσφέρει δυνατότητες ε, να σπουδάσει κανείς στο εξωτερικό και θεωρούμε ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια στενότερη συνεργασία μεταξύ του Εράσμου και του Γιούρες κάτι που θα διευκόλυνε αυτήν την ε, διασυνοριακή κινητικότητα και που με τη σειρά της θα οδηγούσε σε καλύτερη αντιστοίχηση φοιτητών σε ανώτατη εκπαίδευση και με τον αυτόν τον τρόπο να αυξήσει την δική τους απασχολησιμότητα. Όσον αφορά τις πρακτικές ασκήσεις, ισχύει το ίδιο ο συσχετισμός δηλαδή με το πρόγραμμα Εράσμος και όσον αφορά τις ε, ασκήσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και το διαφορετικό ε, ρυθμιστικό καθεστώς που ισχύει σε κάθε κράτος μέλους. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές ε, και μεταξύ των κρατομελών αλλά και σε, εντός των ίδιων κρατών μελών ορισμένες φορές μεταξύ των περιφερειών τους. Άλλες χώρες έχουν ένα πρόγραμμα που βασίζεται περισσότερο στο χώρο εργασία ή άλλες σε προγράμματα που βασίζονται περισσότερο στο εκπαιδευτικό σύστημα και πρέπει να λαμβάνετε υπόψη αυτό. Και μια πιο τεχνική παρατήρηση πώς εμφανίζονται οι πληροφορίες για τις πρακτικές ασκήσεις στο πόρταλ, ιδιαιτερότητα, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, αν πάρει κανείς το, το σύστημα Joule, θα πρέπει να δίνονται συγκεκριμένες πληροφορίες όσον αφορά την συμβατική σχέση που συνάπτει κανείς με τις εταιρείε, ε, πρακτικές ε, πληροφορίες αλλά και ο μισθός. Και ένα τελευταίο σχόλιο αφορά το ρόλο των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων να γνωμοδοτούν επί των εθνικών σχεδίων δράσης. Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται σε εθνικό επίπεδο με τη συμμετοχή των κατάλληλων ε, φορέων. Δεν θεωρούμε ότι οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι δηλαδή θα πρέπει να γνωμοδοτούν επί των εθνικών σχεδίων δράσης στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στην ε, κυρία Ντενάς από την ΕΤΟΚ, την Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε για να συμμετάσχουμε στην ανταλλαγή απόψεων για την ε, πρόταση για τον κανονισμό για το δίκτυο Γιούρες. Εμείς στην Συνομοσπονδία των Συνεργοδημιουργών έχουμε εμπλακεί ε, ενεργά ευθύ εξ αρχή με αυτή την υπόθεση και ακόμα και πριν το 1994 που είχαμε την ε, επίσημη ίδρυση του Γιούρες. Βεβαίω και εμεί θέλουμε την κινητικότητα, αλλά αυτό να γίνεται με δίκαιου όρου και επίση ε, κατά τη δική μα γνώμη η κινητικότητα ε, ακόμα και αν έχει ψηλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η λύση ε, εν του προβλήματος της ανεργία. διότι αν δεν έχουμε θέση απασχόληση ταυτοχρόνω, τότε αυτό είναι μια ψευδέστηση για να το πούμε έτσι οπότε θα πρέπει να δείτε το ότι εμείς ενδιαφερόμαστε, συμφωνούμε και για τις υπηρεσίε του κρατικού τομέα. Επίσης ε, υπάρχει ομοφωνία στο να υπάρξουν τελικά ποιοτικέ θέσει απασχόληση, ακριβώ και αυτά που είπε και ο κύριο Πλάμερ όσον αφορά την κινητικότητα των μαθητευομένων, ε, εκπαιδευομένων και εμεί φυσικά και με όλα αυτά συμφωνούμε, όμω θέλουμε αυτά να γίνονται ε, με δίκαιο τρόπο. Δεν χρειάζεται να μπω στις ε, λεπτομέρειες, ξέρετε τι εννοούμε. Ε, σήμερα δε γνωρίζετε ότι έχουμε πάρα πολύ ευξημένη προτεραιότητα για την κινητικότητα και στην νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναζητούμε την κοινωνική κινητικότητα όσο να από τις δεξιοτήτων και ταυτόχρονα επίσης έχουμε την οδηγία σε σχέση με την εφαρμογή το και υλοποίηση των υπαρχόντων δικαιωμάτων των ε, κυκλοφορούντων ε, εργαζομένων που έχουν την κινητικότητα δηλαδή. Συμφωνούμε και με τις τροπολογίες και με την εφαρμογή του σχεδίου ε, κανονισμού ή και γι' αυτό και θεωρούμε ότι αυτό ε, η δίκαιη αναγνώριση του ότι πρέπει το δίκτυο Γιούρες να το ενισχύσουμε στα πλαίσια αυτής της οδηγίας. Επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο των κοινωνικών εταίρων που είναι πολύ σημαντικός για πληροφόρηση, για παροχή συμβουλών και για εξασφάλιση των δικαιωμάτων των ε, εργαζομένων που έχουν την κινητικότητα. Επίσης, να αναφερθούμε στο ότι η εφαρμοστική οδηγία αφορά τα κράτη-μέλη που θα πρέπει να ανοίξουν κάποιες υπηρεσίες, κάποια γραφεία για να εξασφαλίσουν την δίκαιη κινητικότητα. Επίσης, εδώ πρέπει να διανοηθούν κάποιο ρόλο οι υπάρχοντες φορείς, γιατί δεν έχει νόημα του να έχει κανένας καινούργιες υπηρεσίες, καινούργια γραφεία. Εμείς έχουμε τα γραφεία του Eures και επίσης τα, τα συνδικάτα μας όταν δεν υπάρχει εταιρική σχέση διασυνοριακή. Τώρα για να έρθουμε στο σχέδιο του κανονισμού. Συμφωνούμε. Αναβαθμίζει το ρόλο του δικτύου Γιούρες. Μετά από 20 χρόνια υπήρχε έλλειψη προβολής του έργου του Γιούρες, τι κάνει, τι γίνεται όσον αφορά τις προσφερόμενες εργασίες. Ήταν θέμα και ελέγχου εισαγωγικά για τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στα πλαίσια των υπηρεσιών του δημοσίου. Και επίσης, αυτό το οποίο τώρα μας απασχολεί και μας απασχολεί από την αρχή είναι η εμπλοχή των υπηρεσιών προσφοράς εργασίας του ιδιωτικού τομέα. Και ακόμη και αν έχουμε κάποιο είδους τρόπο ελέγχου της συμμετοχή το πλαίσιο δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο σήμερα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ένα πλαίσιο, ένα πλαίσιο εποπτείας, ελέγχου της συμμετοχής. Στο ίδιο πλαίσιο πρέπει τώρα στα πλαίσια του δικτύου να έχουμε πλήρη εμπλοκή των κοινωνικών εταιρών, όχι μόνο σε επίπεδο ένωσης, αλλά και σε περιφερειακό. Στις διασυνορικές ε, τελικές σχέσεις, όπως είπατε, στα συμβούλια, στην ε, ε, Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ελεύθερη Διακίνηση Εργαζομένων, παντού. υπάρξει και επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωστεί και σε εθνικό επίπεδο των κοινωνικών εταίρων. και να συμμετάσχουν στην Εθνική Υπηρεσία Συντονισμού. Στην ομάδα συντονισμού του Γιούρες ασχοληθήκαμε με αυτό και τι μας είπανε ότι ναι, αναγνωρίζεται το ρόλο των κοινωνικών εταίρων, αλλά ακόμα δεν έχουν το ρόλο που του αρμόζει. Τώρα, κάτι άλλο και σημαντικό είναι η διασυνοριακή εταιρική σχέση. Για μα είναι πάρα πολύ σημαντικό ω ε, ένα φορέα και εκεί εμπλέγονται οι κοινωνικοί εταιρείοι. και εδώ έχουμε κάποιο διαπεριφερειακό συμβούλιο συνδικάτων Μερικές χώρες ε, ακόμα και απαγορεύεται, οπότε δεν πρόκειται για γενικό διάλογο αυθεντικό, αλλά πρόκειται για εταιρική σχέση, για να μπορέσουμε να, ξε, να ε, ανταλλάσσουμε πληροφορίες όσον αφορά το τι κάνουν 18 ε, συμβουλευτικοί φορείς της Eures και Συμβουλή των Εργοδοτών. Όλα αυτά όμω δεν καλύπτονται από τον ε, ε, κανονισμό. Θέλουμε μια απλή μνήμα στη διασυνοριακή συνεργασία. Είχαμε μια έρευνα πάρα πολύ πρόσφατη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει για ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες ε, αλλά μαζί κοντά σε αυτούς είναι και η οικογένειά του κλπ. Οπότε δεν είναι μόνο αυτοί. Εκτό από το θέμα του δικτύου σε 28 κρατη Τόσο το μάλλον καθώ υπάρχουν πολλοί φραγμοί και γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι νέα εμπόδια και φραγμοί αναδύονται, δημιουργούνται και στα πλαίσια θεμάτων κοινωνική πρόνοια, ε, εργατική νομοθεσία και φορολογία. Ακόμα και όταν έχουμε διμερείς συμφωνίες για την φορολογία, πέραν αυτών έχουμε άλλα, άλλα εμπόδια και φραγμούς. Να, τα βασικά μηνύματα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων της ETUC. Ε, Ευχαρίστω να απαντήσω στις τυχόν ερωτήσεις και διευκρινήσεις. Ευχαριστούμε. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Άρκινς, ο οποίος είναι ε, υπεύθυνος του Γιούρες για τις κλαματικές υπηρεσίες απασχόλησης. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας για το θέμα αυτό του Γιούρες που ήδη βρίσκεται επιτάπητος εδώ 14 χρόνια προς τη μεταρρύθμιση του. Αυτά τα τέσσερα χρόνια έχουν αλλάξει πολλά ως προς την ε, κατάσταση και τη διάθεση που επικρατεί στο τραπέζι των δημοτεύσεων. Ε, ενημερωτικά να πω ότι στη δική μας, στη φλαμανδική, στο φλαμανδικό σκέλος, ε, προβλέψαμε την συνιστόσα γιούρες στις υπηρεσίες μας, το ίδιο και για τη διεθνή κινητικότητα, αλλά και την διαπεριφερειακή κινητικότητα. Υπάρχει αλλαγή στη χρήση του γιούρες, ε, με προσφορά πληροφοριών και ε, συμβουλές καθοδήγηση σε όλες τις ε, δράσεις μας στη VDAB, ε, την Φλαμαντική Υπηρεσία Απασχόλησης, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πλήρη στοιχεία, όπως για την πληροφορική, την υγεία, την εργονομία, αλλά αυτά δεν τα φέρνουμε σπερασμόνοι μας. Έχουμε πολλούς ε, συνεργάτες Και αυτό γιατί είμαστε έτσι πιο αποτελεσματικοί, έχουμε περισσότερες γνώσεις, με εμπειρογνώμονες, ενός εμπειρογνωμόνων για τις κατάλληλες πληροφορίες και γι' αυτό το λόγο συνεργαζόμαστε όχι μόνο με τους κοινωνικούς εταίρους αλλά και με τις ιδιωτικές υπηρεσίες ενημέρωσης ή πληροφόρησης. Ως VDAB έχουμε συμφωνία με τις υπηρεσίες απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα περίπου 3.000 τέτοιες υπηρεσίες για να συμπληρώνουμε τα κενά στη βάση δεδομένων μας. Και αυτά τα δεδομένα περνάνε απευθείας και στη βάση δεδομένων γιούρες. Αυτό από το 2012 μας έχει δώσει κάποια πρώτα αποτελέσματα. Με 300 κοινές που έχουν συμπληρωθεί. Μπορεί να πείτε ότι δεν είναι πολλά, αλλά Εάν με ρωτούσατε το 2012 τι θα γινόταν, δεν θα είχα να σας πω τίποτα. Μάλλον μηδέν θα σας έλεγα. Για αυτές λοιπόν τις κοινές θέσεις, μία από τις τέσσερις είναι στον ιδιωτικό τομέα. Ε, η συνεργασία μας λοιπόν ήδη υπάρχει. Και ήδη σε κάποιο βαθμό εφαρμόζουμε αυτή την ιδέα μεταρρύθμισης του Γιούρες και του σχετικού κανονισμού. Στηρίζουμε λοιπόν τις εταιρικές σχέσεις, την κάλυψη των ε, καινούν θέσεων και όπως βλέπει τώρα και η VDAB που μπορεί να χρησιμοποιηθούν και από άλλες υπηρεσίες για την απασχόληση ε, καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι η κατεύθυνση που πρέπει να επιδιώξουμε. Όμως έχουμε ακόμη κάποιες δυσκολίες με τον νέο κανονισμό που προτείνεται. Συμφωνούμε όπως είπα να υπάρχει διαφάνεια στην αγορά εργασίας και κάλυψη των κενών θέσεων. Και να είμαστε βέβαιοι ότι η μετατόπιση από την πληροφόρηση στην αντιστήχηση των πληροφοριών θα οδηγήσει σε ένα στεγνό εργαλείο αντιστήχησης. χρειάζεται ακόμη σοβαρή προσπάθεια σωστή καθοδήγηση και θα πρέπει εδώ να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. επίση να καταπολεμήσουμε το κοινωνικό αποκλεισμό ε, μένοντας πάντοτε στα πλαίσια του Γιούρες, διότι δημόσια κονδύλια ε, είναι αυτά που ε, χειρίζεται αυτό το δίκτυο και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Για τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων είναι σημαντική όχι μόνο για την κοινωνική εταίρεια, αλλά γιατί έχουν μια μεγάλη πείρα στα θέματα αυτά. Εάν λοιπόν θέλουμε να ενημερώσουμε τους ε, ε υπεύθυνου για την αναζήτηση εργασίας ή τους εργοδότες, ε, είναι ήδη κάποιες ιδέες. Για τις πρακτικές ασκήσεις και τις μαθητείες θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε δυσκολίες. Ε, ήδη στο Βέλγιο δοκιμάσαμε και κάποιοι λένε ότι το Βέλγιο είναι και μικροαθία της Ευρώπης. Πραγματικά υποφέραμε. Υποφέραμε για να καταφέρουμε, πώς να το πω, για να μπορέσουμε να το διοργανώσουμε όλο αυτό. Για να καταφέρουμε να έχουμε σωστό σύστημα πρακτικής άσκησης και μαθητείας και εκτός συνόρων μεταξύ των δύο επαρχιών του Βελγίου. Αυτό φανταστείτε να γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τι έχει να συμβεί. Για μας είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε και τον έλεγχο εφαρμοζοντα αυτό τον νέο κανονισμό για το επαγγελματικό ε, άκθος και τον αντίκτυπο μπορεί να έχει. Και για το θέμα της ΕΣΚΟ. Σημαντικό είναι να έχουμε ένα σύστημα που να επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε η ΕΣΚΟ να πάει στη σωστή κατεύθυνση. Είμαι περίεργος γιατί το εργαλείο δεν είναι ακόμη έτοιμο να αναφέρεται στον κανονισμό. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε και γιατί πράγμα θα δεσμευτούμε. Πριν δεσμευτούμε. Είναι πολύ σημαντικό επίση για μας που είμαστε κρατική υπηρεσία απασχόληση να έχουμε συνεργασία με όλου του ομολόγου μα σε όλα τα επίπεδα και να μην υπάρχει υπερβολική ρύθμιση αλλά ευελιξία, διαλεκτικότητα στην υλοποίηση όλων αυτών των μέτρων. θα πρέπει και οι υπηρεσίες για τι αναπασχόλησει στον ιδιωτικό τομέα να έχουν συνεργασία με όλους τους απαραίτητους φορείς, όπως το Γραφείο του Συντονισμού. Εμείς στη VDAB έχουμε συνεργασία με το σχετικό γραφείο, αλλά είμαστε και οι ίδιοι ε, γραφείο συντονισμού. Για να ολοκληρώσω λοιπόν. Ελπίζω να απέδειξα ότι δεν φοβούμαστε να συνεργαστούμε με οποιουσδήποτε ενδιαφερόμενους εδώ και τους συναδέλφους που βρίσκονται στην ίδια στα ίδια έδρανα μαζί μου. Και βεβαίω μπορούμε να βρούμε συμβαστικέ λύσει για τον κανονισμό που προτείνεται, όμω παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ποιε θα είναι οι συνέπειε του κανονισμού εφόσον εφαρμοστεί. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Ο λόγος του κύριο Πένελ, διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρεών Απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση που απευθύνεται στη EuroSet σε αυτήν την άκροση για το EURES που θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της κινητικότητας που πιστεύουμε ότι πρέπει να ενισχυθεί. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στο πώς οι δημόσιες και οι ιδιωτικές ε, υπηρεσίες μπορούν να συνεργαστούν για να στεφθεί το Γιούρες με επιτυχία. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει το Γιούρες να έχει, ε, έχει αμφισβητηθεί το αν θα πρέπει να ε, ανοιχτεί το Γιούρες στους ιδιώτες. Πρώτον νομικά το δικαστήριο θεώρησε ότι η δημοσίευση θέσεων απασχόλησης είναι οικονομική δραστηριότητα και γι' αυτό το λόγο εναντιποτίθεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και ένας επιχειρησιακός λόγος. Όπως γνωρίζετε, οι αγορές εργασίας στην Ευρώπη δεν λειτουργούν τόσο καλά όσο θα έπρεπε και έχουμε περισσότερους από 25 εκατομμύρια πολίτες που ψάχνουν δουλειά και ταυτόχρονα έχουμε εκατομμύρια κενές θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί. Δεν ξέρουμε ακριβώ τον, ε, τον αριθμό αυτών των κοινών θέσεων. Ε, είναι προφανέ πάντω ότι υπάρχει έλλειψη διαφάνεια, έλλειψη αντιστοίχηση στην ε, αγορά εργασία, έλλειψη κινητικότητα των εργαζομένων που μειώνει την δυνατότητα των εργαζομένων που ψάχνουν δουλειά να βρουν δουλειά. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων φορέων και να κοινοτοποιηθούν όλοι οι παράγοντε και οι φορεί για να βρουν οι άνθρωποι δουλειές. Γι' αυτό και η δική μου οργάνωση ε, υποστηρίζει ιδιαίτερα την πλατφόρμα Γιούρες και το άνοιγμα της στους, ε, στις ε, δημόσιες θέσεις απασχόλησης. Το πρόβλημα, το ερώτημα είναι πώς μπορεί να γίνει η καλύτερη αξιοποίηση και από την πλευρά του Γιούρες υπάρχουν διάφορες προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρούνται. Ως γενική αρχή θα λέγαμε ότι η ιδιωτική ιδιωτικές και οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει στο βαθμό του, δυνατό, στο βαθμό του δυνατού να ε, δραστηριοποιούνται επίσης όρις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα βάσει του εγγράφου που συζητούμε. Πρώτα απ' όλα θεωρούμε ότι οι ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει να μπορούν να γίνουν και μέλη και εταίροι του γιούρας για να αποφευθεί η διακριτική μεταχείριση η ιδιότητα του πλήρους μέλους του Γιούρις δεν μπορεί να ε, αποδίδεται μόνο στους δημόσιους φορείς. Το Γιούρις θα πρέπει να είναι μια ε, αρχή που θα περιλαμβάνει και δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης και θα πρέπει να έχει ως στόχο να εκπληρώνει όλα τα καθήκοντα που περιγράφονται στο άρθρο 9 του εγγράφου που συζητούμε. Και αν δεν προσφέρουν όλες αυτές τις ε, υπηρεσίες, τότε θα πρέπει να υπάρχουν εταιρικέ σχέσεις με ιδιωτικούς φόρους. Αυτή η ευελιξία είναι προϋπόθεση για να αυξηθεί και η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα του Γιούρες. Άλλο θέμα είναι πώς θα επιλέγονται οι εταίροι του Eures. Από τη δική μας πλευρά η επιλογή αυτή δεν θα πρέπει να εναποτίθεται μόνο στις εθνικές αρχές. Ακόμα και η έλλειψη πολιτικής βούλησης ε, για να δημιουργηθεί συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε κάποια κράτη-μέλη ενδέχεται να δημιουργήσει συγκρούσεις συμφερόντων. Ξέρετε, από δημόσιες αρχές που επιτρέπουν σε ιδιώτες φορείς να εισέρχονται στο γύρος. Η λύση είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για, να, ε, για το ποιος θα μπορεί να γίνει μέλος του EURUS και αυτό θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και το γεγονός ότι κάποια από τα μέλη θα είναι διεθνείς εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι αν θα, αν θα θέλουν να δημοσιοποιήσουν κάποια κενή θέση τους θα πρέπει να τη δημοσιεύουν και στα 28 κράτη-μέλη και εξετάζοντας το εθνικό επίπεδο το σύστημα διαπίστευσης θα πρέπει να βασίζεται όσον αφορά, ε, όσο το δυνατόν περισσότερο στο υπάρχον σύστημα αδειοδότησης που ε, εφαρμόζεται σε 25 κράτη-μέλη. Και αυτό είναι μια ε, θα πρέπει να, περιλαμβάνει και μια διαδικασία ανάκλησης της ιδιότητας του μήλου σε περίπτωση που υπάρχουν ε, ε, καταγγελίες. Επίσης υπάρχουν τρεις βασικές υπηρεσίες του Γιούρες. Τα βιογραφικά, οι κενές θέσεις και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες. Θα πρέπει τα βιογραφικά να μπορούν να κοινοποιούνται σε ανώνυμη μορφή για την προστασία της ιδιωτικότητας. Γνωρίζετε ότι κάποιες εταιρείες και κάποιοι αναζητούντες εργασία δεν θέλουν να γνωρίζουν, να κοινοποιούνται τα στοιχεία τους στη διαδικασία αυτή. Και τέλος, στο άρθρο 18, παράγραφος 6, για, τις, ε, για τα τέλη που θα χρεώνονται, Θεωρούμε ότι η διάταξη αυτή δεν ευθυγραμμίζεται με, το, με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία διότι αναφέρει ότι τα τέλη δεν θα πρέπει να διακρίνονται μεταξύ των ε, διαφόρων υπηρεσιών. Για μας ε, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη διάταξη έτσι όπως έχει διατυπωθεί στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και σε ό,τι αφορά την συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων θα θέλαμε να πούμε ότι είναι απαραίτητη για τη μεταρρύθμιση του γιούρες αλλά οι προϋποθέσεις που έχουν θεσπιστεί για να γίνει κανείς μέλος του γιούρες νομίζουμε ότι είναι υπερβολικά αυστηρές και ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο τη μεταρρύθμιση του γιούρες. Η οργάνωση που εκπροσωπώ είναι πέρα για πέρα ανοιχτή για να συζητήσουμε ε, τους καλύτερους δυνατούς τρόπους ε, συνεργασίας που έχουμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ πολύ. At, ε, ο Μάρκ, κύριος Χέιντεν. Μαρκ κυριος ο οποίος είναι συντονιστής ε, στην ε, διασυνορική περιφέρεια του Ρήνου και του Μοζέλα για το Euros. Θα σε ευχαριστώ εγώ. Από την πάνω μπορώ να μιλήσω τη γλώσσα μου. Κυρίε και κύριοι, εγώ είμαι ο συντονιστή τη ε, περιοχή Μοζελαρίνου. Στο Γιούρε δεν είναι πολύ μεγάλη αυτή η περιοχή. Να σας πω ακριβώς τι κάνουμε. Ε, αποτελεί μια τέτοια εταιρική σχέση με 50 υπηρεσίες και υπηρεσίες επίσης δημοσιολάβησης Γερμανοί, Ολλανδοί, ε, Βέλγοι σε αυτή την Euroregio όπως λέγεται και εκεί έχουμε μια διεσυνορική συνεργασία αναπτύξη. Επίσης έχουμε και κάποια σημεία ενημερωτικών γραφείων στο Άχεν, στο Μάστριχτ, στο Χάσελ, στην Λιέγη και <clears throat> μιλούμε για εκατοντάδες χιλιάδων διασυνορικών εργαζομένων και 4 εκατομμύρια κατοίκων σε αυτήν την περιοχή. Ε, ξεκινήσαμε λίγο πριν το δίκτυο του Eures το 1993 και επίσης αυτή η εταιρική σχέση υποστηρίζεται από το Eures της περιοχής Μοζελαρίνου. Όσο με τη χρηματοδότηση, η χρηματοδότησή μας προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ...200.000 ευρώ για τις επιδοτήσεις που λάβαμε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Έχουμε δε υποβάλει μια πρόταση για τον πρώτο διαγωνισμό σύμφωνα με όσα ισχύουν από τον, σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης έχουμε προβλέψει κάποιες νέες ε, διαδικασίες ότι μόνο δημόσιες υπηρεσίες μπορούν να υποβάλουν προσφορές. Οπότε άλλα μέχρι τώρα γιατί από τώρα και μέχρι του χρόνου θα ισχύει αυτό που σας είπα νέα διαδικασία. Τώρα να σας περιγράψω πώς έχει αυτή η εταιρική σχέση, να σας πω τι θέματα έχουμε κάθε μέρα να αντιμετωπίσουμε όσον αφορά τις ε, παροχέ μας προς τους πολίτες τις υπηρεσίες. Μπορεί κανεί να πάρει το ποδηλατό του και να περάσει τα σύνορα. Και αυτό δίνει μια καινούργια διάσταση στα πράγματα. Αν κανείς λοιπόν μπορεί να περάσει με το ποδήλατο σε μια άλλη χώρα Αυτό είναι ένα θέμα. Όταν κάποιος όμως είναι διασυνορικός εργαζόμενος μπορεί να το κάνει αυτό μέχρι να πεθάνει. Άρα πρέπει ο κόσμος να ξέρει αυτού του είδους ε, η εργασία ε, στη διασυνορική υφής τι ακριβώς σημαίνει και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την οδηγία για τον συντονισμό των υπηρεσιών κοινωνικής ασφαλίσεως. Αυτό βέβαια μας ξεπερνά γιατί εμείς θέλουμε, έχουμε έναν πυρήνα θέματα που μας απασχολούν γιατί σχεδόν απαγορεύεται να ενημερώνουμε σχετικά με αυτό. Άρα εδώ έχουμε ένα κενό στο νόμο το οποίο θα πρέπει να αρθεί και θα πρέπει να βρούμε προσωπικό το οποίο να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Έχουμε επομένως ε, κάποιους επαγγελματίε, επαγγελματίες, και Χρειάζεται επομένω να μπορούμε να καλύψουμε και την επίλυση διαφορών. Πολλές φορές έχουμε ε, ανάγκη για παροχή συμβουλών, ε, τώρα είναι και οι οικογένειες των εργαζομένων, περιπλέγονται τα πράγματα και αυτό επίσης έχει συνέπειες όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Πέραν του ότι έχουμε και κάποιους ιονίες ε, αυτό αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι είναι δύσκολα εργαζόμενοι. Αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε μέρα και προσπαθούμε να βρούμε απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Πρόσφατα έχουμε μία βελτιωμένη στρατηγική που υιοθετήσαμε Σαν γιατροί είναι οι σύμβουλοι μας. Πρέπει πρώτα να διαγνώσουν το πρόβλημα που τους παρουσιάζεται. Δεν μπορούν να τα κάνουν όλα, μπορούν να τα λύσουν όλα. Ε, αλλά όταν δεν μπορούν, ακριβώ σαν τον ε, παθολόγο, ε, υποδεικνύουν ποιο είναι ο ειδικό που θα λύσει το πρόβλημα. Έχουμε και υπηρεσίες φοροτεχνικές για αντίστοιχε συμβουλές. Πάντα για τους διασυνορικούς εργαζομένους. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες δημιουργήθηκαν και εξελίχθηκαν σε αυτή μας την διαδρομή μες στον χρόνο. Έγινε περισσότερος ο συντονισμός, καλύτερος, ε, διαρθρώθηκε καλύτερη συνεργασία μας δηλαδή και όμως δεν νομίζω ότι λήφθη υπόψη αυτή η πτυχή του θέματος από την προτινωμένη οδηγία. Χάρη στο Κοινοβούλιο. υπάρχει προϋποδότηση. Θετικό αυτό. Και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ε, ε, νομοθεσία σχετική με το EASY σε σχέση με την νομοθεσία για το EURES. Τώρα, εν κατακλείδη, θα σας πω τα εξής τρία. Κοιτάξτε τι γίνεται όσον αφορά την προχή πληροφόρηση σε μια διασυνοριακή ε, περιφέρεια. Δεν είναι θέμα μόνο προσλήψεως εργαζομένων. Είναι το να καλύψουν κάποιες ανάγκες ε, που υπάρχουν διαβίου από αυτούς τους εργαζομένους. Και μέχρι στιγμής δεν τους καλύπτουμε 100%. Στις παραμεθόρες περιοχές είναι σωστό να έχουμε εταιρικέ σχέσεις και αυτό θα πρέπει να γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο επίσης. Διάφορες μορφές ε, συνεργασίας όπως και να συγκροτούνται. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα πρέπει να κάνουν τα κρατημέλη. Και φυσικά πρόκειται για του χαρακτήρα όταν μιλούμε για διασυνοριακά θέματα. Και νομίζω ότι αυτή η νομοθεσία που συζητούμε σήμερα αντικατοπτρίζει αυτά όλα που σα εξήγησε. Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Να δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Χάιντς Πέκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι πυρογνώμονε. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για τις παρεμβάσεις σας και σας ευχαριστώ για αυτό που μας προσφέρατε ήδη από τώρα. Προσωπικά ως, έχω πρόσβαση ως σκιώδης εισηγητής στο δίκτυο που αποφασίστηκε στον τριμερή διάλογο, το δίκτυο των δημόσιων φορέων απασχόλησης στις αρχές του έτους. Και εκεί χαιρέτησα την πρωτοβουλία της Κομισιόν και θεωρώ ότι και εσείς Θεωρείτε θεωρείτε ότι είναι σημαντικό διότι η πλατφόρμα Euros θα πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική και θα πρέπει να ενισχυθούν οι δυνατότητες που προσφέρει το, το Euros. Σωστά σημειώσατε ότι υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ του αριθμού των, των ανέργων και εκείνων που αναζητούν εργασία και ότι υπάρχει ένα πρόβλημα να καλυφθούν και απασχόλησης τις ε, εκτιμήσεις σας και τις θέσεις που εκφράσατε θα ήθελα να μου τις ε, αποστείλετε γιατί θα τις ε, αξιολογήσουμε και στο, στην πορεία των εργασιών μας και θα καταλήξουμε και στο τι από αυτά μπορούμε να υιοθετήσουμε. Πολύ σύντομα να αναφερθώ σε ορισμένα ζητήματα που ενδεχομένως θα μπορέσουν να αποτελέσουν ε, συγκεκριμένα ερωτήματα. Από τα σχόλια αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια αμφιβολία όσον αφορά την συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης. Από την άλλη πλευρά, μάθαμε από το φλαμανδικό πρόγραμμα ότι κάτι τέτοιο μπορεί πολύ καλά να λειτουργήσει. Και γι' αυτόν τον λόγο το ερώτημά μου είναι το εξής. Πώς φαντάζεστε και το ερώτημα απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Συνδικάτων και της ε, Eurocheat. Πώς φαντάζεστε λοιπόν εσείς ότι αυτή η εταιρική σχέση και η ιδιότητα πλήρους μέλους μπορεί με ρεαλιστικούς όρους να απαντηθεί. Γιατί εδώ υπάρχουν διάφορες ερμηνείες, ακούστηκαν πολλές ερμηνείες και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι στο ζήτημα αυτό θα πρέπει να υπάρχει πράγματι μία προτεραιότητα των δημόσιων φορέων, διότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το κίνδυνο του cherry picking. Και επειδή υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να διαλέγει κανείς τι τον Ε, εκείνων που 150.000 και εκείνων των ανθρώπων που είναι διατηθμένοι να μετακινηθούν που ανέρχονται σε 3 εκατομμύρια τότε το πρόβλημα ε, προέρχεται από την ε, διαφήμιση πιστεύετε ότι έχετε επαρκείς πόρους για όλα αυτά που πρέπει να γίνουν δεύτερο ερώτημα Ακούσαμε διάφορα σχόλια από διάφορα ερευνητικά Ινστιτούτα, βάσει των οποίων, παρά το γεγονός ότι οι σύμβολοι του Γιούρες είναι ικανοί και αφοσιωμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, παρόλα αυτά υπάρχει μια ανισότιμη ποιότητα στην, των υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών. Αλλά ορισμένες φορές ακόμη και εντός του ίδιου κράτους μέλους οι ετούντες ε, εργασία λαμβάνουν διαφορετικές πληροφορίες από διαφορετικούς συμβούλους. Έχετε κάποιες συγκεκριμένε προτάσεις για το πώς μπορούν να βελτιωθούν οι υπηρεσίες, η ποιότητα των υπηρεσιών, πώς ε, γίνεται Πώς θα μπορούσαν, για παράδειγμα, οι υπάλληλοι του Γιούρες να λειτουργούν ως γενικοί ιατροί, πώς, ε, στους οποίους θα προσέρχονται οι άνθρωποι που να ζητούν εργασίες ως, προς, ως πρώτος σταθμός. Έχετε κάποιες ιδέες για το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Ευχαριστώ. Έχοντας ακούσει όλες αυτές τις ερωτήσεις, νομίζω ότι δύο μπορούν να απαντήσουν μόνον ο κ. Άτκινς. Ναι, είχαμε και άλλες ερωτήσεις βέβαια. Να τις θέσουμε. Η κυρία Γιασλοβιέσκα. συγχωρείτε που το σκότωσα. Έχω κάποιες ερωτήσεις και θα ήθελα να σας, να σας ζητήσω να τις απαντήσετε. Ποιος είναι ο λόγος που το Γιούρες δεν ενδιαφέρεται για συνεργασία με ιδιωτικού φορείς με τις, ιδιωτικές, με τις υπηρεσίες για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα και η παρακολούθηση όσων βοηθήσατε και διευκολύνατε την εξέπρεση εργασίας. Έχετε κοιτάξει και μελετήσει ποτέ για πόσο καιρό ε, τελικά έχουν απασχόληση αυτοί οι άνθρωποι. Επίσης ποιο είναι το μέσο κόστος, κατά μέσο όρο το κόστος για να βρει ε, μια θέση εργασίας ένα άτομο βάσει των υπηρεσιών που προσφέρετε. Και ποια εργαλεία χρησιμοποιείτε για να είστε αποτελεσματικότεροι. Και έπειτα από δική, σας, από τη δική μου εμπειρία γνωρίζω Γνωρίζω ότι μπορεί να υπάρχει μεγάλη ποικιλία ε, στους τρόπους που μπορεί να εξεύρε κανείς μια θέση εργασίας, ακόμα και με τη δική του πρωτοβουλία. Πώς μπορούμε λοιπόν να κινητοποιήσουμε τους ανθρώπους να κάνουν περισσότερα για να βρουν δουλειά. Εσείς την τελευταία ερώτηση. Και εγώ να σας ευχαριστήσω όλους τους εμπειρογνώμους. Σε αντίθεση με άλλους ομιλητές, νομίζω ότι το Eures είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που χαιρετίστηκε και από τους εμπειρογνώμονες ομόψυχα, αν και υπάρχουν κάποιες ανησυχίες. Δύο ερωτήσεις όμως έχω. Πρώτον, για τις ε, πρακτικές ασκήσεις και τις μαθητείες. Σύμφωνα με την Κομισιόν υπάρχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Ποιος συμμετέχει, έχει ξεκινήσει, υπάρχουν εμπειρίες που ε, θα μπορούσαμε να μαζέψουμε. Δεύτερον, γνωρίζω τις δυσκολίες που αφορούν την ισορροπία μεταξύ δεξιοτήτων, μεταξύ των διαφορών κρατών μελών. Αλλά δεν είναι πλέον υπερόριμο αυτό το ζήτημα. Δεν είναι επιτέλους απαραίτητο να εκδοθούν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές με βάση τις οποίες θα απλοποιηθούν τα θέματα που σχετίζονται με, τα, με την κοινωνική ασφάλιση. Ιδιαίτερα στις διασυνορικές περιοχές νομίζω ότι είναι μια ε, καθημερινή ε, κατάσταση την οποία ε, αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι εκεί. Ναι, ευχαριστώ. Θα έλεγα ότι ε, ελπίζω ότι δύο από εσά θα προσπαθήσουν τουλάχιστον να απαντήσουν στα ερωτήματα. Ο Έρικ Άρκαντ και ο Ντένις Πέναλ και αν υπάρχει και κάποιος άλλος που θεωρεί ότι μπορεί να προσθέσει κάτι, βεβαίως θα το κάνει. Κύριε Άρκενς, εσείς ε, έχετε το λόγο πρώτος. Yes. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω στα Ολλανδικά, αν μου επιτρέπετε. Um, quite a lot of questions here. Uh, sorry. <laughs> Πολλές ερωτήσεις, με συγχωρείτε. Είναι πολλές ερωτήσεις που ε, ακούσαμε. Σε ό,τι αφορά την ε, συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, για τους ιδιωτικούς και δημόσιους μεσολαβητές, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να συνεργαστούμε σε ισότιμη βάση. Γνωρίζω ότι οι σχέσεις μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα δεν είναι ομαλές σε όλα τα κατημέλη ε, για διαφορετικούς λόγους. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος βέβαια για να τους αναπτύξω, αλλά στη Φλάνδρα ε, βλέπω ότι αν ε, ως VDAB τοποθετηθούμε στα θέματα αυτά και προσπαθήσουμε για την αγορά εργασίας να της δώσουμε, ε, να την ε, οδηγήσουμε προσφέροντας πληροφορίες όσους αναζητούν θέση εργασίας, τότε ως VDAB Έχουμε κάνει τεράστιες προσπάθειες για να έχουμε όσο δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες μέσω υπολογιστών κιόλα, που διατίθενται και σε ιδιώτες. Η τράπεζα των δεδομένων μας είναι από τις πλέον επισκέψιμες στην ε, Φλάνδρα. Και βεβαίως τη χρησιμοποιούν και οι ενδιαφερόμενοι από τον ιδιωτικό τομέα μπορούν να αναφερθούν σε αυτές τις θέσεις γιατί κοιτάζουν τη δική μας τράπεζα δεδομένων και παράλληλα έχουν πρόσβαση όσοι αναζητούν δουλειά. Είναι λοιπόν σημαντικό δημόσιος και ιδιωτικός τομέας να ανταλλάξουν υπηρεσίε που οδηγούν στην επίτευξη των κοινών μα στόχων. Παρόλο που είναι λίγο διαφορετική μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Αν μπορούμε όμως να συμφωνήσουμε και να καταλάβουμε ή με τα δικαιώματα των ΔΕ, μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Σε ό,τι αφορά την διάθεση όλων των ε, εργαλείων που διατίθενται, πρέπει να διαπιστώσω ότι η DDB εδώ και χρόνια έχει ακολουθήσει αυτή την πολιτική όλα, ε, όλες οι θέσεις που γνωρίζουμε και που ε, φτάνουν στα χέρια μας ε, δημοσιεύονται στο πόρταλ του Γιούρες. Όμως έτσι όπως, έτσι όπως είναι οργανωμένο σήμερα δεν είναι πολύ εύκολο να το χρησιμοποιούν. Οι ενδιαφερόμενοι ξέρω ότι εργάζεται σκληρά η Επιτροπή αυτή τη στιγμή για να δημιουργήσει τη δυνατότητα, την καλύτερη δυνατή ε, τράπεζα δεδομένων και σε συνεργασία με την ΕΣΚΟ στο μέλλον. Βλέπουμε επίσης και προσπαθούμε να, όπως ρωτήσατε και εσείς, να δούμε αν έχουμε αρκετά μέσα στη διάθεσή μας για να έρθουν όλα αυτά εις πέρας. Όπως είπα και στην αρχική μου εισήγηση, πολλά εξαρτώνται από την υλοποίηση αυτού του κανονισμού. Από το πώς όλα αυτά θα ερμηνευτούν με αυστηρότητα. Περιέχει πολλά στοιχεία ο κανονισμός. Και εμείς ως VDB κάνουμε ό,τι μπορούμε και σε συμφωνία με τον ιδιωτικό τομέα και για την ε, κάλυψη θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει ένα νέο σύστημα που θα επέτρεπε στον ιδιωτικό τομέα πλήρη συμμετοχή. Γιατί στην πράξη κάποιες φορές αυτό είναι απαραίτητο. Τώρα για το πόσο είναι γνωστό το Γιούρες. Ως δημόσιος ε, δημοσιολογητής. έχουμε εμείς την εξής ε, μέθοδο. Εάν κάποιος ψάχνει θέση εργασία πρέπει να ε, βρει δουλειά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ακόμα και ένα στο εξωτερικό που να το στηρίξουμε. Εάν κάποιος είναι στο εξωτερικό, λοιπόν, μπορούμε να βοηθήσουμε. Αλλά Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το Eures, διότι ως VDB έχουμε μία θύμη στην Φλάνδρα και για την διεθνή μας διάσταση. Όποιος ψάχνει δουλειά, οποιοδήποτε προσφέρει δουλειά ε, και τον εξυπηρετήσουμε, τον ευκολύνουμε εμείς, θα σταθεί στο ότι βοηθήθηκε, όχι αν βοηθήθηκε από ένα συγκεκριμένο γραφείο, μια υπηρεσία συμβούλων, γιούρες ή κάτι άλλο. Στα, στις υπηρεσίες της VDVA χρησιμοποιούμε πλήρως το όσα προσφέρει το γιούρες, γιατί η διεθνή συνεργασία είναι ένα μέρος της καθημερινής μας δουλειάς. Κύριε να δω λίγο αν υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις οποίες δεν έχω απαντήσει. Ναι, για, το, για ποιο λόγο το Γιούρες δεν είναι πρόθυμο να δουλέψει με ιδιωτικές εταιρείες. Οφείλεται στις εμπειρίες από κράτη-μέλη. Κάποια κράτη-μέλη δεν έχουν κανένα πρόβλημα με κάτι τέτοιο, αλλά σε άλλα κράτη-μέλη οι άνθρωποι αντιδρούν πάρα πολύ έντονα. Και αυτό που βλέπετε στο κείμενο είναι μια προσπάθεια να συμβιβαστούν αυτές οι δύο εντελώς διαφορετικές θέσεις. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μπορούν να συμμετέχουν οι φορείς ως εταίροι δεν έχουμε πρόβλημα με αυτό, αλλά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τον τρόπο που το κάνουμε, ώστε οι κενές θέσεις από τον ιδιωτικό τομέα να μπορούν να δημοσιοποιούνται στην, στο γιούρες και οι δημόσιες ε, υπηρεσίες απασχόλησης μπορούν να επιτελέσουν το έργο αυτό. Θα προσπαθήσουμε να συμπληρώνουμε τις πληροφορίες που έχουμε ώστε να εξυπηρετούμε την αγορά εργασίας στην Φλάνδρα. Αν υπάρχει κάποιο ερώτημα που ξέχασα, ζητώ συγγνώμη, αλλά υπήρχαν πάρα πολλά θέματα. Ίσως ο Μάρκ Χέντες μπορεί να μας απαντήσει. Είχα και μια ερώτηση από τον κύριο Μαρτάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε πολύ σύντομα απλώς να στηρίξω τα λόγια κάποιων από τους παρεμβαίνοντες προηγουμένως ιδίως των ε, ε, παρεμβαίνοντα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων για το ρόλο που θα πρέπει να έχουν οι κοινωνικοί εταίροι νομίζω ότι σε ορισμένες πλατφόρμες ε, όπως και στην περίπτωση του Γιουρές υπάρχει ένα θέμα διεύθυνσης, διαχείρισης την περασμένη χρονιά ήμουνα στην, στο Τρίερ στη Γερμανία όπου συμμετείχα σε σχετική συνεδρία συνεδρίαση και βλέπουμε ότι εκπροσώποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ανησυχούν. Και νομίζω ότι αυτό είναι αντιφατικό σε σχέση με τα όσα είπαμε προηγουμένω για τη θέση των νέων και την καταπολέμηση τη ανεργία. Πώ θα υπάρξει κινητικότητα εάν δεν έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα εργαλεία για να μειωθεί η ανεργία, ιδίω των νέων. Νομίζω ότι αντιφάσκουμε. Εάν είναι θέμα κόστους, ο νέος που προηγουμένως μας μίλησε για ε, κόστος 150.000 ευρώ από την ενέργεια των νέων, εδώ νομίζω ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε ως προσπάθεια. Κάποιο θα πρέπει να μα απαντήσει, διότι τα υπόλοιπα ε, θα είναι απλώ θέμα τοποθέτηση για ένα διάστημα, αλλά δεν αρκεί αυτό. Εδώ παίζουν τεράστιο ρόλο και κοινωνικοί εταίροι, συμβουλευτικό, ενημερωτικό, γνωρίζουν τι ε, συγκεκριμένε περιοχέ, έχουν γνώσει τοπικού επίπεδου, γνωρίζουν του ηθήνοντε. Το θέμα λοιπόν είναι τι κάνουν ε, με το Γιούρε, τι μπορεί να κάνουν οι συνδικαλιστικέ οργανώσει πώ μπορεί να βοηθήσουν από κοινού όλη την καταπολέμηση τη ανεργία. Can you, να πείτε κάτι σύντομα, κύριε Άρκιν. Ευχαριστώ. Όσον αφορά αυτές τις δαπάνες και το κόστος ως VDB συνεργόμαστε με τα συνδικάτα και υποστηρίζεται οικονομικά αυτή η συνεργασία όποτε υπάρξει ανάγκη. Δεν ξέρω πώς μπορεί να σας καλύψει ε, πληρέστερα συνάδελφος από τα συνδικάτα τι γίνεται σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε χώρα γιατί Προσπαθούμε να έχουμε όσο γίνεται πιο άρτια συνεργασία σε επίπεδο γιούρες. Να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομη, να σας τα πω στα γαλλικά για αυτό το λόγο. Après, je reviendrai sur RES, au rôle... Euh, αυτό που είπατε πρώτα-πρώτα για τον, τον βασικό ρόλο του, του τη συνεργασία μεταξύ των ε, δημοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών. Και τι γίνεται όσον αφορά το τέλος του μονοπωλίου του δημοσίου. Αυτό έχει γίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Με ε, κάποια απόφαση του Γραφείου εργασία. Αυτό είναι το πάγιο επιχείρημα. Εδώ και 10 χρόνια. Οπότε εμείς συμφωνούμε πλέον δεν έχουμε επιλογή. Άπαξ και υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία τηρούνται. Άπαξ και έχουμε την απόφαση του Γιούρες, υπάρχει μια συγγραφή υποχρεώσεων που αφορά αυτές τις ιδιωτικές ε, εταιρείε. Τηρούν τα όσα επιτάσσει το Γιούρες. Και όποτε έχουμε τίποτε εκτροπές ασχολούμεθα με αυτά τα φαινόμενα όπου υπάρχει τέλος πάντων επίσης παράδοση σε κάποια χώρη ε, ιδιωτικών εταιριών. Υπάρχει επομένω αυτό το είδους πλαισίωση που ισχύει. Είτε έχουμε επομένως συντονισμό του γιούρες και επίσης ε, έχουμε και εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων. Είχαμε επομένως κάποιο είδους ε, παρεκβάσεις και εκτροπές κάπου μεταξύ Γαλλίας και Καταλωνίας. Εκεί ε, είχε γίνει κάποια κίνηση για την Ανδόρα, κάποια συγχώνευση τέλος πάντων υπηρεσιών. Και είπαμε ότι λόγω της συμμετοχής των συνδικάτων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προχώρησε το θέμα, γιατί είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της όσον αφορά το πόσο όλα αυτά θα περιχαρακωθούν. Κατάλαβα τι λέει ο κύριος Βουλευτής για την προσφορά εργασίας με τυχή αμοιβή και τι γίνεται με τη βάση δεδομένων. Αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να διαβεβαιώσουμε ότι κάποια κρατημέλη πλέον δεν παίζουν με τους όρους αυτούς του παιχνιδιού και πια δεν είναι το γιούρες το οποίο ανακατεύεται και δεν θέλουν πλέον να φροντίσουν την κινητικότητα. Ε, ή φοβούνται τη φύγη των εγκεφάλων κλπ. Σα το λέω, γιατί εδώ και 20 χρόνια ασχολούμαι με τον συντονισμό των δικτύων. Θα το πούν και οι συνάδελφοι. Οπότε πολλές φορές λέει το αρμόδιο Υπουργείο θα κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς για την γεννητικότητα. Και έτσι προχωράνε κάποια κρατημέλη. Αυτό μην το ξεχνάμε, θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Επίσης, είναι αλήθεια ότι η παρακολούθηση των προσφορών εργασία για κάποιους λόγους, λόγους των κρατικών αρχών, δεν γίνεται πλήρως. Και εδώ πάλι θα πρέπει να αναμειχθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως γίνεται. Οπότε έχουμε κάποιες προσφορές που μπαίνουν, μπαίνουν στο παιχνίδι από τις, από εταιρείε. Και αυτό κάπως νοθεύει, μπερδεύει το πράγμα όσον αφορά την ποιότητα της απασχόλησης. Να επανέλθω πάντως συγκεκριμένα στο τι γίνεται τώρα όσον αφορά τις συνέπειες της χρηματοοικονομικής κρίσης και τι γίνεται με το αποτέλεσμα της απόρριψης των ε, ε, διασυνεργαζομένων. Δηλαδή για το ότι τους αρνούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά τη σχέση με την ε, χώρα προελεύσης, την επιστροφή τους. Μιλούμε τώρα για δύο εκατομμύρια προσώπων που θέλουν να μετακινηθούν, θέλουν να πάνε να δουλέψουν αλλού. Και υπάρχει βέβαια και αυτό το φαινόμενο της ε, απόρριψης τους διώχνουν κάποιες χώρες ε, όπως το Βέλγιο και η Μεγάλη Βρετανία. Τώρα παρακολουθούμε την κατάσταση από κοντά και παρακολουθούμε πού γίνεται αυτό, ο κόσμος δεν θα πάει όπου να είναι. Πρέπει να έχουμε να πάνε στα, στα γραφεία πληροφόρησης, στα γραφεία γύρω στις ε, περιοχές. Και σε κάποιες χώρες τα πράγματα μπερδεύονται ακόμη παραπάνω. Σε κάποιους ε, ευρωπόλους Ε, και κοντά στο Λουξεμβούργο και εκεί που πρέπει να επισημαίνεται το πρόβλημα να λύνεται πολλές φορές εκεί επιτόπου αλλά ο στόχος μας είναι να υπάρχει λύση γενική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως αυτό το σχέδιο κανονισμού η πρόεδρος διακόπτη συγγνώμη αλλά έχουμε άλλα δύο λεπτά διερμηνίας και έχουμε ακόμα ένα θέμα στη μέση Πρέπει να σας διακόψω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, το γιούρες δηλαδή, αλλά θα επανέλθουμε. Δεν θα αποφασίσουμε χωρίς να ακούσουμε τα πάντα. Ακούσαμε πολλά σήμερα το απόγευμα και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας. Θα πρέπει να συζητήσουμε το τελευταίο θέμα της μεσαίας διατάξεως. Γιατί πολύ σύντομα δεν θα έχουμε διερμηνία. Thank you very much for all your contributions. Uh, our last uh, uh, point on the agenda, the European Investment Bank, the annual report 2013. Για την ετήσια έκθεση για την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρότεινα όσο λιγότερο γίνεται να παρέμβουν για ένα λεπτό μόνο οι διερμηνείς να μην μέχρι να τελειώσουμε. Question. Ερώτημα. Δεν μπορούμε να αναβάλουμε το θέμα αυτό για την επόμενη συνεδρίαση. Όχι, δεν μπορούμε, λέει η Πρόεδρος. Πρέπει να αποφασίσουμε σήμερα για αυτό το θέμα. Ναι. one minute. Κύριε Λόπες, ένα λεπτό. Κύριε Λόπε, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να σα μιλήσω πάρα πολύ σύντομα και να σα εξηγήσω τι πέντε βασικέ τάσει των ε, τροπολογιών μια που δεν έχουμε χρόνο. Νομίζουμε ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία να σας πω ότι έχει σημασία για μας πρώτα πρώτα δεν μπορεί να υπάρχει μια τόσο συντηρητική ε, πολιτική από την ΕΤΕ για τις ε, επενδύσεις θέλουμε και ιδιωτικά καλά θέλουμε για τα, για τριπλά α να συνεχίσουμε και έτσι να έχουμε στην ε, Ευρώπη απασχόληση. Δεύτερον, θα πρέπει να έχουμε περιβαλλοντική αξιολόγηση και κοινωνική όσον αφορά τα προγράμματα. Να υποστηριχθεί δηλαδή η ποιότητα τρίτων να υπάρχει μια διαχείριση πιο δημοκρατική στην τράπεζα και υπάρχει ε, μεγάλο περιθώριο βελτίωσης αυτό. Να εστιαστούν οι προσπάθειες στην απασχόληση, την ποιοτική, καλύτερη συμμετοχή των γυναικών, μείωση της ανεργίας της μακροπρόθεσμης και έτσι να ευνοηθούν και οι πιο ευάλωτες κοινωνία. Όλοι τα δεσμικά όργανα έχουν ένα ρόλο να παίξουν σε όλα αυτά και επίσης σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντική και αυτό θέλουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει να λάβουμε υπόψη το, το, ψηφιακό, τους ε, ανθρωπίνους ε, πόρους κλπ. Για να μπορούσαμε να καλύψουμε αυτό, το χαμηλό στα τελευταίο, των τελευταίων ετών. Κύριε Ευχαριστώ. 30 δευτερόλεπτα. Πρώτα-πρώτα, αν υπομονώ να έχουμε καλή συνεργασία με τον κύριο Κάζα. Είμαι βεβαίω ότι αυτό θα συμβεί. Οι τροπολογίε που έχω αποβάλει για την κοινωνική οικονομία, τις δημοσιονομικές λύσεις για τα μέλη. Μπορούμε να βρούμε, πιστεύω, τις κατάλληλες λύσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και άλλοι συνάδελφοι όπως ο Τόμας Μάν έχουν πολύ καλές τροπολογίες εδώ. Είμαι σίγουρο ότι θα φτάσουμε, όπως είπα, σε ένα αίσιο πέρας. Και καλή συμφωνία. Ευχαριστώ. Mr. Rowling. Oui, un peu très rapidement. Ο κύριος Ζολά, ε, ευχαριστώ πολύ σύντομα. Κύριος Κάζα, σας ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Γι' αυτό ζήτησε να διαβάσω εγώ τις απόψεις του. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις 60 τροπολογίες που υποβλήθηκαν. Να πω ότι μια σειρά από τις τροπολογίες θα γίνουν δεκτές, ιδίως αυτές που προσθέτουν ε, τις ε, κατάλληλες πληροφορίες από στατιστικής πλευράς και αυτές που στοχεύουν στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή εκείνες που θέλουν να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Επίσης αυτές που ζητούν λιγότερη ρύθμιση και περισσότερη ευελιξία στη διαχείριση των κοντιλίων της ΕΤΕ. Αντιθέτως ο κύριος Τιάζα δεν θέλει να, να δεχτεί τις τροπολογίες που δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στο δημόσιο τομέα και τη δημιουργία τη από αυτόν, και να μην δημιουργηθούν περιτά εμπόδια στην ΕΤΕΠ. Είναι σαφές ότι όλα αυτά τα στοιχεία ο κύριος Κάζα ως εισηγητής θα έχει τη χαρά να τα συζητήσει για να βρούμε συμβαστικές λύσεις με τους διάφορους και όντις εισηγητές τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, δεν έχουμε χρόνο παρότι είναι σημαντική η έκθεση αυτή, αλλά διαπίστωσα ότι λόγω των πολλών τροπολογιών κινούμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Θα πρέπει να δοθούν περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να επιφέρουμε αποτελέσματα. Στις συζητήσεις με τους κοιόδους νομίζω ότι το θέμα 10 είναι σημαντικό. Μιλάμε εκεί για μια νέα δομημένη διαδικασία επικοινωνίας. Την τελευταία εβδομάδα στο Στρασβούργο ζήσαμε, βιώσαμε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ήταν ε, μια ευκαιρία ο κύριος Χόιερ, ε, ο πρόεδρος ε, της Τράπεζας Επενδύσεων, να μιλήσει στο Κοινοβούλιο. Και είναι μια πολύ καλή προσέγγιση αυτή θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια. Είναι πρόθυμη και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για κάτι τέτοιο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει δομημένη διαδικασία. Δεν θα πρέπει να είναι απλά μια, μια τράπεζα που θα έχει την έδρα της στο Λουξεμβούργο, αλλά θα πρέπει να είναι μια τράπεζα που θα μπορεί να επιφέρει πραγματικά αποτελέσματα και θα ήθελα να καλέσω όλους να συμμετέχουν σε αυτήν την νέα διαδικασία. Νομίζω ότι θα ήταν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για όλους. Ευχαριστώ κύριο Μπάλας. Ευχαριστώ. Να πω το θέμα της διαφάνειας είναι καθοριστικής σημασία. Θα πρέπει να ζητήσουμε και το Συμβούλιο και η Επιτροπή να λάβουν κάποιο ρόλο, κυρίως με όσα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή προτείνονται από τον κύριο ε, Γιούνκερ. Τώρα, εμείς ως Κοινοβούλιο δεν πρέπει και στο επίπεδο τη ΕΤΕ να κάνουμε κάποιε προτάσει. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο δημοκρατικό έλεγχο, ακόμη και εκεί για να παίξουμε το ρόλο μας ως ε, βουλευτέ. Και για τις δράσεις της ΕΤΕ θα πρέπει να έχουμε ε, οπωσδήποτε ενημέρωση διαρκώ, ιδίω για να ξέρουμε τι χρηματοδοτεί στα περιβαλλοντικά και ιδίω ε, υπό το φως του σχεδίου Γιούνκερ όπως προτάθηκε. Αυτά τα τρία στοιχεία ήθελα να παρατηρήσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Χρυσεντεύσκη. Τα πολωνικά, ελπίζω. Πρόεδρε, Ευχαριστώ. Να πω ότι κατά την άποψή μου και για την δική μας την ομάδα, του συντηρητικού και μεταρρυθμιστές, αυτό το κείμενο είναι μια καλή βάση για να έχουμε μια κοινή θέση με τροπολογίες. Συνάδελφοι, νομίζω συμφωνούμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πρέπει να βρούμε και νέα χρηματοδοτικά μέσα. Όμως να επιμείνω σε μία πτυχή θα πρέπει να μας απασχολήσει το μέλλον της τράπεζας που καλό θα είναι να προσφέρει ε, δημοσιονομικά μέσα λαμβάνοντας και τις ανάγκες χωρών με αγορές κεφαλαίων ή ε, ανάγκες λιγότερο αναπτυγμένες. Θα μπορούσε να είναι και μέσα η εργαλεία απλά στη χρήση, αλλά να μπορούν και τα κράτη αυτά να έχουν πρόσβαση στις πιστώσεις, κάτι πως τώρα δεν ε, ήταν ε, δυνατό σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπό το φως αυτών προσπαθούμε να Υποβάλλουμε κάποιες τροπολογίες. Πρόεδρος, ήταν ε, κουραστική και μακρά η μέρα μας. Ε, τελικά δεν ήταν καλός όμως ο προγραμματισμός. Όταν φτάσαμε στο Γιούρες δεν ήξερα ότι θα πάρει τόσο χρόνο και ενέργεια. Όμως ευχαριστώ όλες και όλους για τις συμβολές τους. Το χρονοδιάγραμμα για την ε, ΕΤΕ και την ετήσια έκθεσή της είναι έγκριση στην Επιτροπή Απασχόλησης 21 και 22 Ιανουαρίου και τότε θα επανέλθουμε και θα συνεδριάσουμε τη νέα χρονιά. Αυτή ήταν η τελευταία μας συνεδρίαση πριν το τέλος της χρονιάς, λίγες εβδομάδες πριν. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μείνατε τόσες πολλές ώρες μαζί μας σήμερα. Για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε όλα τα θέματα που πρέπει να ολοκληρωθούν σήμερα. Ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε και τους διερμηνείς.